Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας. Παρακαλώ καθίστε. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι από ό,τι βλέπω. Ε, υπάρχει και μετάδοση διαδικτυακά. Και διερμηνία έχουμε σε 20 γλώσσες με εξαίρεση αστονικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και γοεδελικά και ελπικά. Γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι ο αντιπρόεδρος μας ο κύριος Βοητσεχόφσκι, τέος πλέον αντιπρόεδρος, εξελέγει μέλος του ελεκτικού συνεδρίου από τις 7 Μαΐου έμεινε και είναι η χειρή θέση του, οπότε θα πρέπει να εκλέξουμε τον αντικαταστάτη του, ε, αντιπρόεδρο δηλαδή, στην Επιτροπή μας. Όπως ξέρετε, εδώ ισχύει το σύστημα DONT. Ο κύριος Βοτσεχόφσκι ήταν από την ομάδα ECR των συντηρητικών μεταρρυθμιστών και άρα αυτή η ομάδα δικαιούται να ορίσει τον υποψηφιό της που θα μας το παρουσιάσει γιατί έχουμε απαρτία οπότε πληρείται αυτή η προϋπόθεση και να διαβάσω τους αναπληρωτές, τα αναπληρωματικά μέλη που αντικαθιστούν εδώ τακτικά μέλη. Σράιερ, ο κύριος Σάντος, Ντανανό, Όζουκ, Βυσνιεύσκα και Χόιμπους είναι οι αναπληρωτές που θα λάβουν μέρος στην ψηφοφορία για την εκλογή του Αντιπροέδρου. Παρακαλώ το συντονιστή τον κύριο Νίκολσον να μας παρουσιάσει την υποψηφιότητα της ομάδας ECR για τη θέση του Αντιπροέδρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που υπάρχει εδώ απαρτία στην έναρξη μιας πολύ σημαντικής συνεδρίας. Εσείς δεν είχαμε στο παρελθόν απαρτία. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς ε, λυπόμαστε ε, που ο προκάτοχος αυτής της θέσης έχει πάρει μια, ένα νέο διορισμό στο συλλεκτικό συνέδριο. Ε, ο κύριος Κίσμεκ είναι αυτός που προτείνουμε, ο οποίος ε, ήταν μέλος του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για πάρα πολλά χρόνια και θέλαμε αυτόν να προτείνουμε ως αντιπρόεδρο για την Επιτροπή Γεωργίας. Ο κύριος Κούσμουκ λοιπόν είναι η υποψηφιότητά μας. Σας ευχαριστώ. Συμφωνία, ο κύριος Κουσμιούκ ε, με την υποψηφιότητά του. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγινιος ζήτησε το λόγο. Είναι περισσότερο ελπίδα παρά προσδοκία. Πριν από δύο χρόνια, αν είχαμε παρακολουθήσει, ακολουθήσει τις παραδόσεις του Κοινοβουλίου η ομάδα η e ε, των, των φιλελεύθερων δημοκρατών θα είχε τώρα έναν αντιπρόεδρο. Όμως ε, δυστυχώς ε, δεν ακολουθήσαμε την παράδοση και το ECR πήρε αυτή τη θέση. Απλώς ήθελα να τονίσω αυτό το ιστορικό στοιχείο για τα αρχεία, Πρόεδρε. Το σημειώνουμε κύριε Άγγινιο. Θα το γράψουμε στα πρακτικά το σχόλιο σας. Θυμόμαστε την κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστούμε για την υπενθύμηση. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε μία υποψηφιότητα έχουμε μόνο, αυτή του κυρίου Κούσμιουκ. Οπότε προτείνω να ψηφίσουμε διαβοής με χειροκρότημα. Ε, δεν υπάρχουν ψήφοι κατά. Πρέπει για το, για το τυπικό να το ρωτήσω. Ούτε αποχές. Κύριε Άγγνιο, ζητήστε το λόγο. Όχι. Δεν είπατε ποιο ψηφίζει κατά. Γι' αυτό σήκωσα το χέρι. Ψηφίζω κατά. Α, μάλιστα. Εντάξει, εντάξει. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Κούσμιου, παρακαλώ ελάτε στο Προεδρείο για να λάβετε τη θέση σας. Ή θέλετε το λόγο, ναι, προτιμώ να μείνω στη θέση μου προς το παρόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια και τον κύριο Νίκολσον, αλλά και τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων, τα μέλη της Επιτροπής μας, γιατί έγινε σεβαστή η αρχή που υιοθετήσαμε κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής μας θητείας, ώστε η οι πολιτικές ομάδες ε, να λαμβάνουν θέσεις. Ε, με την αποχώρησή του ο κύριος ε, Βοητσεχόφσκι άφησε μία θέση κενή την οποία δικαιούται να πληρώσει η ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Έγινε σεβαστή αυτή η αρχή και σας ευχαριστώ θερμά. Επίσης, θα ήθελα να δηλώσω ότι θα συνεχίσω το έργο μου σε αυτή την Επιτροπή. Είμαι ταυτόχρονα βέβαια μέλος και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, το γνωρίζετε, γιατί θα έχουμε και την διάμεση αναθεώρηση και βλέπουμε τι απόπειρε γίνονται να αφαιρεθούν, να περικοπούν κονδύλια από το γεωργικό προϋπολογισμό. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι ως μέλος ε, της Επιτροπής Γεωργίας θα μεταφέρω τα σχόλια της Επιτροπής Γεωργίας ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και από αυτή την άποψη θα ε, είμαι πολύ χρήσιμος νομίζω για την ανάπτυξη γεωργίας και για την προάσπιση των γεωργών. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Βουλευτά. Ελάτε παρακαλώ στο Προεδρείο να λάβετε τη θέση σας του Αντιπροέδρου. Είναι όντως σημαντική αυτή η περίοδος που εξετάζουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Η κυρία Μόη ζήτησε το λόγο. Κυρία Μόη, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ. Απλώ ήθελα να τονίσω κάτι για να διασφαλίσω ότι είναι ξεκάθαρο. Στην αρχή της θητείας ήμουν υποψήφιος αντιπρόεδρος αλλά με το σύστημα don't, ε, αυτό που τότε διακηρύσατε, για πρώτη φορά δεν έγινε σεβαστό στη δική μου περίπτωση και εγώ προσωπικά ε, ήμουν υποψήφια για αντιπρόεδρος. Δεν μου φαίνεται λοιπόν δίκαιο κάποιες φορές να διακηρύσουμε τον κανόνα Ντεόντ όταν βολεύει κάποιες ομάδες και όταν δεν σας βολεύει να το ξεχνάμε και να παρεμποδίζονται υποψηφιότητες ε, κάποιων ε, υποψηφίων, μάλιστα απροκάλυπτα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φερά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σημειωθεί στα πρακτικά ότι ο κύριος Φεράν και εγώ δεν θα θέλαμε να λάβουμε μέρος στην ψηφοφορία. Δεν χρειάζεται να σημειώνουμε τι αρνητικέ ψήφου, γιατί η ψηφοφορία γίνεται διαβόη. Ο κύριο Νίκολσον. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επιμακρύνω τη συζήτηση, να μακρηγορήσω, αλλά να με σαφείς. Η θέση του Προέδρου των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών υπέρ του κανόνα Ντεόντ δεν σημαίνει ότι προσπαθήσαμε να σφετριστούμε τη θέση κάποιου. Θέλω να το ξεκαθαρίσω σε όσου ε, κάνουν σχετικά σχόλια σήμερα. Μην κατηγορείτε του ε, συντηρητικού και μεταρρύθμιστε για όλα αυτά. Δική σα άποψη βέβαια, αλλά. Ο κύριο Σάγκνη γελάει, αλλά να μην ξεχνάει ότι ανέκαθεν προσπιζόταν το κανοναντεόν τη ομάδα Αυτό κάναμε πάντα και λυπάμαι λίγο που προσπαθήσατε να κλέψετε λίγο από την υποψηφιότητα του κ. Κιούσμακ με την Προεδρία της Επιτροπής Γεωργίας. Ο κύριος Κούσμακ είναι άξιος υποψήφιος και θα τα πάει πολύ καλά πιστεύω να αναλάβει. Οπότε είναι έγκυρη υποψηφιότητά του. Μάλιστα. Μια και δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο, επαναλαμβάνοντα τα συγχαρητήριά μα προ τον εκλεγέντα αντιπρόεδρό μα, τον κύριο Κούσμιουκ. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, την έγκριση των πρακτικών τη τη 14 14η και 15η Μαρτίου του 2016. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, δεν βλέπω παρατηρήσεις, οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Ένα-δύο λεπτά διάλειμμα μέχρι ότου έρθει ο Επίτροπος Χόγκαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξη που προβλέπει την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τον Επίτροπο Χόγκαν όπως ξέρετε, ο διαρθρωμένος διάλογος προβλέπεται στα πλαίσια της Διοργανικής Συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Και γίνεται το πρώτο εξάμεινο του καθέτους μεταξύ της ε, αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και του αρμόδιου Επιτρόπου. Οπότε έχουμε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο με βάση την ανάλυση των αναγκών και από νομοθετική και μη νομοθετική άποψη. Ε, μάλιστα θα μας βοηθήσει αυτή η συζήτηση για να επιλέξουμε μια σειρά προτεραιοτήτων ε, που θα πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017, αλλά ταυτόχρονα θα κάνουμε και μια αξιολόγηση του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016. Έχουμε μάλιστα και πρόσωπο της ε, Ολλανδικής Προεδρίας ε, και έχουμε μετά τη Σλοβακική. Είναι σημαντική αυτή η εποχή που διανύουμε, οπότε είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο στα πλαίσια αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου που είναι απαραίτητος. Και άλλωστε Έχουμε τακτικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως με τον Επίτροπο που είναι πρόθυμος και έρχεται κάθε φορά που τον προσκαλούμε και τον ευχαριστούμε θερμά για τη στάση του αυτή. Μάλιστα αυτή η οικονομική συζήτηση για τη Γεωργία είναι απαραίτητη. Και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτος αυτός ο διάλογος. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Χόγκαν και κατόπιν Στου συντονιστέ. Παρακαλώ κύριε που έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας για τη δεύτερη φάση του διορθωμένου μα διαλόγου. Έχουμε μια πολύτιμη ευκαιρία να έχουμε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και βάσει του προγράμματος εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017. Έχει περάσει σχεδόν ένα χρόνο, ε, σχεδόν ένας χρόνος από τον πρώτη φάση του διορθωμένου μας διαλόγου και ξέρουμε ότι ήταν ε, χρονιά δύσκολη για τους γεωργούς μας, ιδίως για αυτούς του χείριου κρέατος και των γαλακτοκομικών, οι οποίοι έχουν ε, σοβαρά προβλήματα. Η κατάσταση της αγοράς και οι χαμηλές τιμές για τους γεωργούς και τους κοινοτρόφους είναι στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού. Και βεβαίω αυτό αφορά όλου του τομεί δραστηριότητα του οποίου έχουμε εμπλοκεί. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε την κρίση στην Γεωργία μαζί σα. Και την επόμενη και μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει και άλλος γύρος ε, συζήτησης για την κρίση των γαλλικών μεγαλακτοπαραγωγικών. Θα το συζητήσουμε και στην Ολομέλεια. Θα ήθελα βέβαια να σας παρουσιάσω μια συνοπτική εικόνα για όλες τις δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε και στις αναρκτήριες παρατηρήσεις μου θα επικεντρωθώ όντω στον γαλακτοκομικό τομέα και τον τομέα του χείριου. Η συνολική διατροφική αλυσίδα έχει βγάλει δυσκολίε και ασκεί πίεση στις τιμές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διεθνή αγορά. Οι εξαγωγέ δημιουργούν ανασφάλεια στην αγορά γενικώ. Είναι δύσκολο να βρεθεί σωστή ισορροπία ακόμα μεταξύ ζήτηση και προσφορά. Υπάρχουν λίγε δυνατότητε για αύξηση τη ε, ζήτηση και δεν φαίνεται να διευθύνεται το θέμα. 5,6% έχει πέσει η παραγωγή γαλακτοκομικών του πρώτο δίμηνο τη φετινή χρονιά σε σχέση με το 2015. Οι κάτω χώρε, 33.000 τόνου, η Γερμανία το ίδιο, 140.000 τόνου η Πολωνία και 130.000 η Ιρλανδία. Περιμέναμε αύξηση στην ε, γαλακτοπαραγωγή τον Μάρτιο κατά 5%. Αλλά λόγω της βαρύτητας της κατάστασης βλέπουμε ότι οι εξαγωγές μας στα γαλακτοκομικά στην αρχή τη χρονιάς ήταν κάπως καλύτερες. Είδαμε οι συνολικέ εξαγωγέ σε αντίστοιχα γάλακτος να αυξάνονται κατά 10%. Με ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις, 123% στο γάλα, 40% ε, στο τυρί και ε, το γάλα ζεσκόνο 4%. Όλοι οι βασικοί μας προορισμοί ως το Φεβρουάριο του 2016, μεταξύ των οποίων και οι ΙΠΑ, αυξήθηκαν κατά 9% ενώ υπήρξε διπλασιασμό των εισαγωγών από την Κίνα. Κάτι που επιβεβαιώνει την ανάκαμψη και την ανάκαμψη αγοραστικής δύναμης της Κίνα ως προς τα γαλακτοκομικά. Ω προ τον χείριο, τον τομέα του χείριου κρέατο, υπήρχαν σοβαρότατε συνέπειε και είδαμε του πρώτου μήνε τη φετινή χρονιά να υπάρχουν κάποια δείγματα Μείωση τη παραγωγή 2,4 λιγότερων σφαγιαστών χείρων στην αρχή τη χρονιά. Η τιμή του χείρου παραμένει βέβαια σταθερή, παρά τα χαμηλά επίπεδα, και η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπεράσει τα 130 ευρώ ε, ανατόνο. Φέτο. Ε, παρά το 60% κρέατο που αποθηκεύσαμε πέρσι το Γενάρη. Αυτά επανήλθαν στην αγορά. Έτσι λοιπόν, παρά τι μεγάλε πιέσει στην αγορά, έχουμε μεγάλε δυσκολίε με τι εξαγωγέ. Οι Αμερικανοί δεν έχουν ακόμα ε, βοηθήσει να βρεθεί σωστή ισορροπία. Τον Φεβρουάριο είδαμε να αυξάνεται κατά 20%. Κατά 26% ο όγκο και 19% η αξία των εισαγωγών να σχέση με το Φεβρουάριο του 2015. Θα ξέρετε τώρα ποια είναι η βασική απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κρίση στη Γεωργία. Ε, ε, ανακοίνωσε 900 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Αλληλεγγύης προς τα κράτη-μέλη απευθείας. Τα κράτη-μέλη μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα έχουν 35 μέρες στη διάθεσή τους για να δαπανίσουν αυτά τα ποσά. Μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα τα κράτη-μέλη είχαν ε, ε, δαπανίσει μόνο το 56% του ποσού αυτού. Έχουμε λοιπόν 235 εκατομμύρια από τα 900 ε, που έχουν μείνει εξόδευτα από το Σεπτέμβριο. Τα 500 που έχουν μείνει αχρησιμοποιείται ως τώρα. Το 2015 όμως είχαν ε, ήδη ξεπεράσει το 90% του ποσού τους σχεδιατροφής. Να μιλήσω για το θέμα των παρεμβάσεων. 190 ε, τόνοι οροφή για το γάλα σε σκόνη ήταν η ε, επιχείρηση που έχουμε οργανώσει στις 19 Απριλίου. Υπήρχε σταθερή τιμή και τιμή παρέμβαση. 25.000 τόνοι αγοράστηκαν επιπλέον ε, για την παρέμβαση. Όμω μέχρι τι 20 Απριλίου σταθερή τιμή οδήγησε σε διπλασιασμό τη οροφή με γοργή αύξηση στην πρόσληψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει προφανώς και περαιτέρω αύξηση στο ανώτερο όριο. Το τελικό μέτρο για το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι το 222 για τη ΣΚΟΑ, που επιτρέπουν ε, στου γεωργού και κτηνοτρόφου ε, εθελοντικέ συμφωνίε για την παραγωγή γάλακτο. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν ευρέω με 85% της συνολικής γαλακτοπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να ωφεληθεί από αυτήν την συμφωνία, από τέτοιου συμφωνίες παρά τους περιορισμούς ε, στην παραγωγή γάλακτος που έχουμε προβλέψει με το άρθρο 222. Αυτά προβλέπονται για διάρκεια εξαμήνου από τις 20 Οκτωβρίου 2016 και θα μπορούσαν να επεκταθούν και για ένα περαιτέρω εξάμεινο. Είναι ένα εθελούσιο εργαλείο, όπως είπαμε, είναι στα χέρια των παραγωγών αποφασίζουν να συμμετάσχουν. Και έχω συναντήσει εκπροσώπους ε, γαλακτοπαραγωγών της Ευρώπης, συνεταιρισμών επίσης, και θα τα ξανασυζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα για να δούμε τι δυνατότητε υπάρχουν. Υπό αυτή την άποψη, θέλω να σα επενέσω, Πρόεδρε, για την διοργάνωση των εκφράσεων αύριο το βράδυ, για να δούμε τι μορφή θα πάρουν όλα αυτά και τι αποτελέσματα ελπίζουμε να έχουν. Ελπίζω να καταλάβουμε καλύτερα τα μέτρα και τι δυνατότητε που προσφέρουν. Και να μην υποτιμηθούν ε, όλα αυτά στο εύρο του. Να μην επιτρέπουν στα κατεμένα να διπλασιάσουν τι κρατικέ βοήθειε και μόνο το χρήμα να κινητοποιεί του παραγωγού να χρησιμοποιήσουν αυτά τα επικοδομητικά μέτρα, μόνο αν το επιθυμούν. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου, Πρόεδρε, θέλω να επικεντρωθώ και στην απλούστευση. Είναι μεγάλη προτεραιότητα η πρώτη πλούστευση τη ΚΑΠ. Υπάρχουν πολλέ προτάσει περί απλούστευση, οι οποίε έρχαν σχεδόν από το 2015, όπω η αποσυνδεδεμένη βοήθεια εθελοντικό, οι αποσυνδεδεμένε βοήθειε, οι νέοι γεωργή, η πρόσβαση στι ε, οργανώσει γεωργών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το χειριστούν ε, οι μηχανισμοί τη διοικητική δίκηση στο κάθε κράτο μέλου. Η ε, κατεξοδότηση πράξη του ΑΙΑΚ ε, κρίθηκε πέρσι τον ε, Μάιο και υπάρχει και το, διαδικασία της κίτρινης κάρτας για τους παραβάτες και για τις δηλώσεις τους, εφόσον οι αιτήσει δεν είναι σωστές για κάποιες ενισχύσεις. Η δημοσίευση και η θέση σε ισχύ κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών θα επιτρέψει να γίνουν πληρωμές μέσα στο 2016 για τα ποσά που δεν έχουν αξιωθεί ακόμα. Ελπίζω να έχω τη στήριξή σα για αυτή τη διαδικασία. Οι δημόσιε διαβουλεύσει για την πρώτη φάση του πρασινίσματο έχει ολοκληρωθεί με 140.000 ενδιαφερόμενου. Ε, οι περισσότερε αιτήσει προέρχονται απευθεία από του γεωργού. Πέραν αυτών των πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλο Ιουνίου θα ετοιμάσει ένα έγγραφο εργασία για την αποτίμηση τη όλη κατάσταση και για τι συνέπειε του πρασινίσματο, καθώ και για τον ίσο κανόνα παιχνιδιών στι δυνατότητε παραγωγή. Η αναθεώρηση αυτή θα ε, συνοδευτεί από αναθεώρηση των άμεσων πληρωμών του πρασινίσματο και τεχνικέ λεπτομέρειε στου εφαρμοστικού κανονισμού. Η απομάκρυνση ε, των ε, διάφορων ε, δυσλειτουργικών κανόνων, ελπίζουμε ότι θα φέρει περιβαλλοντικά ωφέλη και μέσα από την όλη διαδικασία του πρασινίσματο, με στόχο να υπάρχει περισσότερη σαφήνεια του τι απαιτείται από του γεωργού και από τι ε, διοικητικέ αρχέ, για να υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερα ωφέλη περιβαλλοντικά και κλιματολογικά από το πρασίνισμα. Οι υπηρεσίε μου επιδιώκουν μια, ε, φιλόδοξη, ένα φιλόδοξο θεματολόγιο προτεραιοτήτων για την απλούστευση, με ίσου κανόνε ε, για όλε τι διοργανώσει ΚΟΑ από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε 150 πράξει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του ε, σχετικού κανονισμού που θα αναθεωρηθούν. Ελπίζουμε τουλάχιστον 20 ε, εφαρμοστικέ και 20 εκτελεστικέ πράξει να έχουν εγκριθεί στο τέλο Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την αναπτύξη τη υπαίθρου τέλο, η διόρθωση τη εφαρμοστική πράξη που εγκρίθηκε στι 20 Απριλίου και ήδη ισχύει θα απλουστεύσει τι ε, υποχρεώσει δημοσίευση για του μικρότερου γεωργού και τι απαιτήσει για την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι θα υπάρχει και λιγότερο άρθρο για τι δημόσιε διοικήσει. Θυμίζω ότι η διόρθωση των χρηματοδοτικών εργαλείων ω μέρο του προγράμματο ανάπτυξη τη υπαίθρου τη Ευρώπη μπορεί να επιτύχει πέραν τη κλασική απλούστευση στα κράτη-μέλη και ενίσχυση για τα περιφερειακά προγράμματα. Στα πλαίσια του προγράμματο εργασία τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη προσπαθούμε να εντείνουμε τι προσπάθειε απλούστευση μέχρι το τέλο τη χρονιά ε, σε ό,τι αφορά τι εφαρμοστικέ και κατεξοδότηση πράξει. Πρόεδρε, έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εγώ για τι εμπορικέ μα διαπραγματεύσει όπω και τα μέλη τη Επιτροπή σα. Δυστυχώ ο τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων για το TTIP τον Απρίλιο δεν έφερε αποτελέσματα και υπάρχει έλλειψη προόδου ω προ τα ευρωπαϊκά συμφέροντα για τα θέματα που αγγίζουν και άπτονται τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε συνεχίζουν να αμφισβητούν ε, του διαπραγματευτικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι γεωργικέ ενδείξει και δεν θέλουν να συμπεριληφθούν τέτοιε διατάξει στην ε, συμφωνία θέλουν την διαγραφή των ημιγενώσιμων ονομασιών ε, για τους γεωργούς, κάτι που προκαλεί αισθήματα ματέωση και απογοήτευσης και από τις δύο πλευρές. Δεν θα περάσω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ε, ιδιαίτερα φιλόδοξη. Θέλουμε να συμφωνήσουμε για ένα, μέτρο, για ένα πακέτο μέτρων φυτογενομικής προστασίας ενισχυμένο στα πλαίσια της συμφωνίας TTIP. Δεν θέλουμε να αποδεχτούμε ένα light, μια light συμφωνία TTIP. αλλά θέλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην ουσία και όχι στην γρήγορη ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η γεωργία και η κτηνοτροφία μα γνωρίζει σοβαρέ κρίσει σε πολλού τομεί και έχουμε και άλλες φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες επιτάπητος ε, όπω την ε, κάλυψη της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στη Συμφωνία Τίτη. Ξέρετε ότι στις 11 Μαΐου ε, αναθεωρήσαμε και την προσφορά μας προς τη Μερκοσούρ ε, για τις ποσοστώσεις του βόηου για τις, και του κρέατος από, την, από τον Μερκοσούρ. αναθεωρήσαμε τις ε, σχετικέ διατάξει και η περαιτέρω αναθεώρηση τη όλη συμφωνία και τη προσφορά μα προ το Μερκοσούρ θα φτάσει τον, στα χέρια μα τον Ιούλιο. Είναι καθοριστική σημασία σε τι τις για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Η διαθεσμική διαδικασία και οι σχετικέ συμφωνίε βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλωσορίζω την δέσμευση τη Προεδρία να επιτύχουμε περαιτέρω πρόεδρο σε αυτού του καθοριστικού τομεί πολιτική και να επιδιώξουμε συμφωνία αυτόν τον Ιούνιο του 2016 για τη βιολογική γεωργία. Εδώ λοιπόν καλωσορίζω το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να είναι φάνταστη και να καλύψει το κενό μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ο μόνιμο εισηγητή, ο κ. Χάουσλινγκ, ε, προσπαθεί να είναι διαλεκτικό και ελπίζουμε ότι όντω θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα και διμερώ να βρούμε λύσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Σα ευχαριστώ για αυτό. Καλωσορίζω την πρόσφατη υπόσχεση και των τριών θεσμικών οργάνων να προσπαθήσουν να επιταχύνουν την συχνότητα οργάνωση τριμερών διαλόγων γιατί ξέρουμε ότι είναι λίγα τα μείζωνα ζητήματα τα οποία παραμένουν εκκρεμή. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμφωνία στο δυνατόν γρηγορότερα. Πρόεδρε, νομίζω ότι κάλυψα μερικά από τα βασικά ζητήματα. Είμαι σίγουρο ότι θα υπάρχουν ερωτήσει που θα ανακύψουν κι άλλα, αλλά στο λίγο χρόνο που μου αναλογεί, ελπίζω ότι μπόρεσα λίγα ζητήματα να τα αναπτύξω τουλάχιστον αρκετά και ελπίζω ότι ήταν επίκαιρα σε προηγούμενε συνεδριάσει σας και παραμένουν επίκαιρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ για την εισαγωγή και σίγουρα στην πορεία της συζήτησης ε, θα ανακύψουν και άλλα σήμερα και θα έχετε την ευκαιρία να σχολιάσετε και να δώσετε απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Περνάμε τώρα στους συντονιστές. Πρώτος ο κύριος Άλμπερτ Ντες. Τρία λεπτά στους συντονιστές. Τρία λεπτά και τίποτα παραπάνω, το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε που είστε εδώ στον διαρθρωμένο διάλογο για δεύτερη φορά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας παρακολουθούσαμε ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρον. Μιλήσατε για την ανισορροπία στην αγορά στο χείριο κρέας και σε άλλα αγροτικά προϊόντα. Επίσης, ε, ε, εγώ ανησυχώ για μια άλλη ανισορροπία είναι η σχέση στην αγορά της ε, εφοδιαστικής αλυσίδας, εμπορικής αλυσίδας. Ε, είχαμε πει ότι θα υπάρξει μια ισορροπία, αλλά βλέπω ότι στην τριμερή διάλογο ε, υπάρχει μια κατάχρηση αυτής της σχέσης ισχύω και δεν μπορούμε αυτό να το αποδεχτούμε στο Κοινοβούλιο να υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι οι οποίοι ε, ε, ας πούμε εμπλέκονται στο επίπεδο της Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν όταν χρειαζόμαστε, όταν έχουμε κάποιες αμφισβητούμενες ε, συμφωνίες είμαστε σκεπτικιστές απέναντί τους. Χρειαζόμαστε 50% γάλα στις συνατορισμούς και 50% στους ιδιώτες ε, αν, ε, δίνετε πάρα πολύ στους, ε, αν, δεν δίνεται πολύ στους μένα χαίρονται οι δε και το ανάποδο. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο χειρισμών και αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, το αναγνωρίζω, θα έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε κατά πόσο ε, σε μια τόσο ισχυρή κρίση ε, στην Ευρώπη θα μπορούσε ένας κανονισμός ε, να μας βοηθήσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να καταστήσουν δυνατό να υπάρχει διπλασιασμός των κρατικών μέτρων. Τα κράτη-μέλη τώρα πρέπει να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Μιλήσατε για την απλοποίηση επίσης ως μέλος του Ευρωκοινοβούλου. Ε, έχω ακούσει πάρα πολλά τέτοια ζητήματα απλούστευσης από την Κομισιόν. Θα ήθελα πραγματικά εδώ να υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια, να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ε, όπως είπατε, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, πολλοί δυσανασχετούν και ε, και όταν μιλάμε για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, ε, όταν γίνονται τροπολογίες και πρέπει να τις αποσύρουμε, ε, υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω επίσης ότι ε, αν κατατεθούν προσπάθειες απλούστευσης και για την TTIP, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το συμφέρον της Ευρώπης στην Γεωργία, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Χόγκαν που είναι και πάλι μαζί μας. Όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν περνάει τις καλύτερες στιγμές της. Οι τιμές είναι χαμηλές σε πολλούς τομείς. Όχι μόνο στο γαλακτοκομικό τομέα και τον τομέα του τύρου. Είναι και πάλι σαφής η ιδιοποίηση των ε, πολιτικών από τα εθνικά κράτη. Βλέπουμε πως οι ΚΟΑ μετατρέπονται σε διανομή ε, πόρων στα κράτη-μέλη, κονδύλια, ε, τα οποία δεν φαίνεται να είναι και αποτελεσματικά. Πολλέ φορέ μάλιστα χρησιμοποιούνται προκαλώντα τα αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκαμε. Εμεί θέλαμε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερε ευρωπαϊκέ αποφάσει για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα στην αγορά και όχι μεμονωμένε αποφάσει των κρατών μελών. Επίση πρέπει να ξανασκεφτούμε ποια είναι τα περιβαλλοντικά ωφέλη του greening, του πρασινίσματο. Με ικανοποίηση χαιρετήσαμε στο Κοινοβούλιο αυτή την ανθεώρηση τη ΚΑΠ την πρόσφατη μεταρρύθμιση τη. Όμως περισσότερα από πνευματικά ωφέλη είδαμε να υπάρχει αύξηση του γραφειοκρατικού άχθου και ο κίνδυνος να προκληθούν περαιτέρω δυσκολίε στα κατημέλη ως προς την ε, εφαρμογή. Εμείς θέλαμε ένα greening πιο ε, εύκολο και εύχριστο και αποτελεσματικό στο, από, από την πλευρά του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών ωφελών, με περισσότερα μετρήσιμα αποτελέσματα και μείωση του γραφειοκρατικού άθου για τα κράτη-μέλη και τις δημόσιες δικήσεις τους. Αυτό επιβάλλεται. Επιβάλλεται αναθεώρηση των ε, εργαλείων αντιμετώπισης των κρίσεων. όπω ξέρετε, Επίτροπε, δοκιμάσαμε στην περασμένη θητεία να προβλέψουμε μέσα πιο ε, εύχριστα για την αντιμετώπιση της διακύμανσης των τιμών και των διάφορων κρίσεων, όμως δεν ε, εισακούστηκαν οι προτάσεις μας, παρέμειναν νεκρό γράμμα. Είναι τρει αυτοί οι σημαντικοί άξονε, γύρω από του οποίου πρέπει να οργανωθεί μια σοβαρή συζήτηση για τη μεταρρύθμιση, την ενδιάμεση αναθεώρηση τη όλη μα ε, προσπάθεια. Το είχαμε πει και από την προηγούμενη θητεία. Χρειάζεται περισσότερη αποτελεσματικότητα στο greening, στο πρασίνισμα, με εργαλεία απαλλαγή από τη γραφειοκρατία και απλούστευση, με μεγαλύτερη έμφαση στην διαχείριση των κρίσεων και με μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο για την Ευρώπη την ίδια. Και γι' αυτό σας ρωτώ για μια ακόμα φορά, Επίτροπε, έχουμε επιτέλου τη δυνατότητα να προβλέψουμε μια ενδιάμεση αναθεώρηση μέχρι τα τέλη του χρόνου ώστε να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τα ενία και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ε, περνάει ο κόσμος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σας ευχαριστώ κύριε Σνίκολσον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ρωτήσω τον ε, Επίτροπο τι διάλογο έχετε με τα κράτη-μέλη σας και το επιτελείο σας σε ό,τι αφορά τις περιοχές ε, ε, με δυσκολίες ιδιαίτερα στο θέμα της γαλακτοπαραγωγής. Γιατί βλέποντας το χάρτη των περιοχών, των περιφερειών αυτών, φοβάμαι ότι οι μηχανισμοί που, και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν ε, καλύπτουν ε, κατάλληλα αυτές τις περιφέρειες. Μάλιστα, ήδη φέτος έχουμε 5% αύξηση της γαλακτοπαραγωγής και αυτό με φοβίζει, με τρομάζει. Είναι πολύ τρομακτική αυτή η κατάσταση και θα πρέπει να περάσει το μήνυμα στην γεωργική κοινότητα και στους ενδιαφερομένους. Γιατί αν συνεχίσουν οι γεωργοί την παραγωγή τους με αυτούς τους ρυθμούς αμύωτους, η κατάσταση ε, δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο και απευκταίο. Ξέρετε ότι στην έκθεσή μου ανέφερα την πρόταση για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για το, γάλακτος, για το γάλα. Είστε υπέρ αυτή τη πρότασης του παρατηρητηρίου γάλακτος. Ε, θεωρείτε ότι θα βοηθήσει την παρακολούθηση της κατάστασης ε, στο γαλακτοκομικό τομέα. Επίσης, πότε θα γίνουν οι ενημερώσεις και η υποβολή εκθέσεων για τα θέματα αυτά. Γιατί περιμένουμε τις εκθέσεις ε, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή την υπερπαραγωγή γάλακτος το συντομότερο δυνατό. Χαίρομαι για τη δήλωσή σας για τις διαπραγματεύσεις στο TTIP. Γιατί ε, φοβόμασταν ότι θα παραμείνουν σημειωτών οι διαπραγματεύσεις ε, του TTIP ε, λόγω των επικείμενων αμερικανικών εκλογών. Αντίθετα, τι γίνεται με το Μερκοσούρ. Η κυρία Μάλστρομ ε, ήταν σαφής γιατί θέλω να μας τα πείτε και εσείς ε, με μεγαλύτερη σαφήνεια. Γιατί πριν από δύο εβδομάδες που μιλήσαμε στο Στρασβούργο φαίνεται ότι πιέζει η κυρία Μάλστρομ για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ. Πιστεύω όμως ότι αν δεν έχουμε αποδείξεις και τεκμήρια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίες και να απορροφούμε τρόφιμα που θα εισάγονται στην Ευρώπη όταν οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι μα είναι τόσο πιεσμένοι και ουσιαστικά ε, πολλούν σε τιμές κόστους. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να απορροφούμε τρόφιμα εισαγόμενα αν δεν αλλάξει κάτι. Τι γίνεται λοιπόν με τις εμπορικές συμφωνίες. Ο κύριος Ρόντε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, παρέμβαση. Κύριε Επίτροπε, ο διαρθρωμένος διάλογος είναι πάντοτε σημαντικός, όμως ε, να σας θυμίσω ότι ο διάλογος είναι πάντοτε μια διμερής μορφή επικοινωνία. Ελπίζω να το καταδείσετε αυτό ε, σήμερα, όχι όπως την τελευταία φορά. Παρατηρήσαμε όλοι ότι αναλαμβάνεται δράση για την κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών και του χοιρινού. Να συμφωνήσω με τον Πάολο όμως, γιατί πραγματικά η πραγματική απειλή είναι η επανεθνικοποίηση του γεωργικού τομέα στην Ευρώπη η ευελιξία μεταξύ των διαφόρων πυλώνων στην ουσία οδηγεί σε αυτή την επανεθνικοποίηση και δεν ναι, ναι, έχουμε ισότιμους όρους ε, για όλους τους αγρότες στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, η πρόταση για τα αέρια του ε, θερμοκηπίου να κάνει το ίδιο. Η ερώτησή μου λοιπόν έχει ως εξής. Θα φτιάξετε μια γενική ανάλυση κινδύνου ε, σχετικά με τις ε, περαιτέρω επανεθνικοποιήσεις ε, στον γεωργικό τομέα συνολικά. Μπορείτε να καταθέσετε προτάσεις για το πώς μπορούμε να προλάβουμε κάτι τέτοιο, όπως ας πούμε μια εγγύηση ότι νέος, ο νέος κανονισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου θα εξασφαλίζει ίσους όρους για όλους και θα έχει και αποτελεσματικότητα σε επίπεδο κόστους ωφέλους. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μας έρχεστε δεν είναι ότι μας φαίνεται κάτι καινούριο. Όλο γύρω από τα ίδια πράγματα τριγυρίζουμε. Περιμέναμε προτάσεις ε, για να λύσουμε την την κρίση που ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Γεωργία, αλλά δεν βλέπω καμία τέτοια πρόταση. Έχω λοιπόν τέσσερις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Στη Γαλλικία, στην πατρίδα μου, οι επιχειρήσεις γαλακτοπαραγωγής καθορίζουν την τιμή του γάλακτο κάνοντας κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους. Αυτό είναι ένα τυποποιημένο αδίκημα με βάση το δίκαιο του ανταγωνισμού. Τι πρόκειται να κάνετε για την κατάσταση αυτή. Επίση, στη Γαλλία 2.244 αιτήσει στήριξη για βιονεκτικές ζώνες και εκτατική κτηνοτροφία απορρίφθησαν εξαιτία των περικοπών και τη πολιτική λιτότητα. Πρόκειται να λάβετε κάποιο μέτρο για να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Ερώτηση τρίτη. Τελευταία, άρχισαν να φαίνονται οι πραγματικές προθέσεις πίσω από τις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Ε, φαίνεται ότι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Γεωργίας ε, στο κοινοτικό ΕΠ μειώνεται κατά 0,8% για το TTIP. Τι πρόκειται να κάνετε. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι θα είναι ευνοϊκή η συμφωνία TTIP για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Επίσης, ε, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις στη ΤΥΠ ε, η μελλοντική εισαγωγή μοσχαρίσιου κρέατος ε, για ένα τομέα που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είσαστε εδώ. Ξέρετε και εσείς ότι γενικά το αίσθημα μεταξύ των γεωργών έχει φτάσει ε, στα, τα επίπεδα και θέλουν να δούνε τι θα γίνει με αυτή την κρίση από την πλευρά των, της Κομισιόν και πότε θα ανακάψουν οι τιμές. Υπάρχει ελπίδα όμως οι γεωργοί δεν θεωρούν ότι μπορεί η Κομισιόν τελικά να κάνει κάτι για αυτό το θέμα. Είπατε ότι καλά πάνε οι εξαγωγές, όμως δεν πάνε καλές γιατί οι αγρότες τελικά δεν παίρνουν καλές τιμές. Είναι η νίκη όταν ε, τελικά δεν αυξάνονται οι τιμές. Ε, αν λοιπόν ε, ακολουθούμε τη λογική ότι μόνο, μόνο ότι οι περισσότερες εξαγωγές είναι καλές, θα πρέπει να κοιτάμε και πώς έρχονται αυτές οι εξαγωγές στην Ευρώπη. Πρέπει να αποφύγουμε η ζήτηση και η προσφορά στην Ευρώπη να μην αντιστοιχούν. Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη ε, να έχουν όλα τα κράτη-μέλη μια μείωση στις ε, ποσότητες γάλακτος, όμως αυτό λέτε ότι θέλετε να το αποφύγετε. Ε, μιλήσατε και για άλλα προγράμματα που όλα σχετίζονται με επιπτώσεις, όμως αυτά ε, δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε γιατί τα, οι αγρότες δεν χρειάζονται περισσότερα, χρήματα, ε, περισσότερα χρέη μέσα από τα χρήματα που θα πάρουν. Οι, οι τράπεζες δεν δίνουν ούτως ή άλλως χρήματα στους γεωργούς πλέον. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών στην γεωργική πολιτική, αλλιώς ε, η κρίση θα παραμείνει και θα έχουμε πολύ μεγάλη μεγάλο πρόβλημα και με τις τιμές. Για το Mercosur επίσης αναφερθήκατε, η κυρία Μάλστρομ ε, κάπως διαφορετικά ακούγεται από ότι εσείς ε, που είναι Επίτροπος Εμπορίου. Έχει ε, πολλές φορές υμνήσει αυτή την συμφωνία, την TTIP. Όμως εμείς ε, μέσα από αυτά που λέει Greenpeace βλέπουμε ότι η TTIP είναι κάτι διαφορετικό. Ε, φαίνεται ότι παίζονται πολλά παιχνίδια κατά της γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να δει αν πρέπει να, γίνει, ε, να προχωρήσουμε εκεί. Και αν πούμε όχι στην TTIP, ε, γιατί να μην γίνει το ίδιο με τη Mercosur. Αν μιλάμε για απελευθέρωση των αγορών, θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η απελευθέρωση. Και κάτι τελευταίο. Το είπαμε ήδη ότι έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση. Ε, έχουμε τη Μονσάντο ε, που τώρα θα την καταπιεί η Μπάγερ. Έχουμε τεράστιους ομίλους γεωργικών προϊόντων. Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση λοιπόν και ε, έχουμε λιγότερους ομίλους, τεράστιους ομίλους που έχουν την εμπορία των σπόρων στην Ευρώπη. Αυτό ε, δεν νομίζω ότι θα είναι καλό ε, και θα συμφωνήσει σίγουρα ο Επίτροπος Ανταγωνισμού για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριος Άγνιου. Είναι πολύ ευχαριστώ να σας ξαναβλέπουμε ε, επιτροπές. Σας είδα και πριν από ένα δεκαπενθήμερο Ε, δεν ήταν τόσο ευχάριστη συγκυρία, αλλά περιμένω και τα σχόλια του κυρίου Φλάναγκαν, διότι θα ενισχύσει τι δικέ μου πολιτικέ απόψει, πιστεύω. Ήμουν προσφάτω σε μία συνάντηση για τη γλυφοσάτη και το κατά πόσον θα απαγορευτεί η χρήση της ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ε, ανθρώπινης υγείας, ε, κινδύνους από καρκίνο ε, και θα δούμε αν αυτό θα συμβεί. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε τρόφιμα από αλλού από την Ευρωπα... εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εισάγουμε και χρησιμοποιούμε άνετα γλυφοσάτη. Ε, έχουμε εισάγει πρόσφατα σπόρους σόγιας που έχουν παραχθεί με τη χρήση αυτής. Κάπου διάβασα ότι η Γαλλία μονομερός θα απαγορεύσει την γλυφοσάτη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο κύριε Επίτροπε. Ένα το μέλο θα ακολουθήσει δική του πολιτική πορεία στη Γεωργία. Μπορεί να απαγορεύσει και την εισαγωγή ε, τροφίμων από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε όπου έχει χρησιμοποιηθεί γλυφοσάτη, λόγω χάρη. Η Γαλλία. Αρχίζει να γίνεται πολύ μπερδεμένο το τοπίο εδώ. Και πραγματικά θα εκτιμούσα τι απόψει σα σχετικά. Επίσης να επισημάνω ότι όσο ε, σχολιάσατε και το θέμα του TTIP είπατε για στόχους. Είναι ασυνήθιστη κατάσταση. Η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να είναι ελεύθερη. Να είναι ελευθερές βοσκής ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίθετο. Ε, στην Ευρώπη λοιπόν ενώ είναι ελευθέρας βοσκής ε, ένα αυγό ε, με συγκεκριμένο ορισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχει λευκό κέλυφος και να είναι και πλημμένο. είναι δύο διαφορετικόμενες, δύο τελείως αντιπαρατηθέμενες απόψεις αυτές. Ποιος θα νικήσει αυτή τη μάχη στη Μεγάλη Βρετανία η θέση μας δεν λαμβάνεται καν υπόψη σε αυτές τις Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε το γύρο με τις ερωτήσεις των συντονιστών. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Ξέχασα τον κύριο Λουαζό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ογκάν, ε, μας λέγατε πέρσι ότι το θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας δεν ήταν δική σας αρμοδιότητα. αλλά δεν φαίνεται να έχετε δώσει σωστή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, διότι αυτό κατέστρεψε και προκάλεσε τόσε βλαβερέ συνέπειε για τη γεωργία μα, κύριε Επίτροπε. Πού είναι η λογική με αθέμετες κυρώσεις, παράλογες που έχουν οδηγήσει σε ασφυξία την αγορά μας, κύριε Επίτροπε, ενώ ταυτόχρονα διαπραγματεύεται τη Διατλαντική Συμφωνία που μπορεί και αυτή να δημιουργήσει προβλήματα στην Ευρώπη. Μην ε, επεκφεύγετε των ευθυνών σα και απαντήστε μου. Και σε ό,τι αφορά την απλούστευση τη ΚΑΠ, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από του μείζονε στόχου και για την ε, εξάσκηση των αρμοδιοτήτων σας ως Επιτρόπου. Αλλά σκέφτεστε τι θα γίνει με τους ε, αδιάκοπους ελέγχους που υφίστανται οι δικοί μας Ευρωπαίοι Γεωργοί και με φόβο να υποβληθούν κυρώσεις είναι οι ελεγκτές ε, ικανοί, είναι αμερόληπτοι, γνωρίζουν καλά τους κανόνες της κάψας. Ειλικρινώς επιζητάτε απλώς πρακτικές λύσεις, διότι εγώ δεν έχω αυτή την εντύπωση. Για παράδειγμα, η θέσπιση προθεσμίας 14-15 ημερών για τους γεωργούς ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν είναι μια καλή λύση. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά τεράστια προσπάθεια κύριε Χόγκαν, είναι κατά από τα μάτια σας ε, οι λύσεις, κατά τη μύτη σας μάλλον και πολλές φορές είναι και προφανείς. Και για την ε, συμφωνία ότι θα είναι αντίθετα με τα συμφέροντά μας. Ε, γιατί συνεχίζετε τις διαπραγματεύσεις. Κατανόητο. Και όσο αφορά το πρασίνισμα, το greening, Ξέρετε τι επιπλέον κόστος θα επιφέρει αυτό για τους ε, παραγωγούς μας και τους γεωργούς μας. Ξέρετε ότι οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές θεωρούνται δυσβάσταχτες, ε, επιβάλλουν επιπλέον φόρτο στους ε, γεωργούς. Και έχουμε ένα τεράστιο αριθμό απαιτήσεων. Νομίζω ότι αν τις αυξήσουμε κι άλλο θα υπάρξουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τρίτες χώρες. Γιατί λοιπόν, γιατί τέτοια αιμονή με αυτή την πολιτική του πρασινίσματος. Ευχαριστώ. Ωραία, τώρα μπορούμε να ξαναδώσουμε το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει μετά τις ερωτήσεις των συντονιστών. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς για την απλοποίηση. Μίλησα για 23 αλλαγέ πέρυσι. Μέσω της απλοποίησης αυτής θα έχουμε ωφέλη για τους ε, αγρότες. Και εφιστώ την προσοχή σας σε αυτές, γιατί θα είναι πολύ χρήσιμες. Καταρχάς, ε, ένας ε, προληπτικός, προκαταρκτικός έλεγχος ε, πριν τις πληρωμές τους αγρότες εισήχθη πέρυσι και μετά από πολλά λάθη που παρατηρήθηκαν, έχουμε την ευκαιρία να τα διορθώνουμε πριν μπουν στα μηχανογραφημένα συστήματα. Άρα, δεν θέλουμε με, αυτό το, θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε το κλίμα φόβου που υπάρχει σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τους επιτόπου ελέγχους. Αν λοιπόν γίνει σωστά η δουλειά με το πνεύμα που εγώ λέω ε, και αυτό περιμένω ότι θα γίνει, ε, τα πράγματα θα πάνε καλά. Ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τα χρήματα κάθε φορά να παίρνουν συμβούλους για να ε, βάζουν σε μια ροή το βασικό τους εισόδημα. Επίσης εξετάσαμε και τους 200 κανονισμούς για τη ΚΟΑ και θα μειώσουμε κατά πολύ το νούμερο αυτό, θα πάμε περίπου στους 40, έτσι ώστε να έχουμε και για τις εθνικές διοικήσεις και για τις ε, φορείς ε, διαχείρισης ε, και λειτουργίας καλύτερη απλούστευση. Μετά, στο πρασίνισμα, στο greening, έχουμε κάνει μια αξιολόγηση, ζητήσαμε τις προτάσεις πολλών μερών για το τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, Είχαμε 3.300 ε, υποβολές προτάσεων στην Κομισιόν, 80% ήταν από αγρότες. Βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο λοιπόν τι συμβαίνει. Θα προτείνω λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες 15 ε, με 20 αλλαγές, ε, τις οποίες πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσουμε για να διαλευκάνουμε την κατάσταση και να μειώσουμε την μη αναγκαία γραφειοκρατία γύρω από την ερμηνεία των πραγμάτων. Ε, θα βελτιώσουμε όπου μπορούμε το περιβαλλοντικό όφελο επίσης ε, που είναι η κεντρική αρχή ε, που περιλαμβάνεται στην νομοθετική διαδικασία για το 2013. Επίσης έχει ο κόσμος ε, λίγο μπερδευτεί, τι γίνεται με τους φράχτες και γενικά όλα τα ζητήματα χωροταξίας είναι ένα θέμα ε, βιοπικιλομορφίας ε, και πρέπει να το προωθήσουμε γιατί αν μειώσουμε την γραφειοκρατία θα έχουμε όφελος για το περιβάλλον. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Δεκάστρο για τα εργαλεία διαχείρισης κινδύου, να πω ότι υπάρχουν τέτοια εργαλεία στην ε, ε, νομοθεσία που έχουμε, αλλά υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στον τομέα και το ε, τεστ της αγοράς που ανέφερε ο κύριος Νίκολσον είναι ένας τρόπος να βελτιώσουμε τα εφιστάμενα μέτρα και κανόνες, αλλά είναι και ένας τρόπος να δούμε και εκτός Ευρώπης, να δούμε τι πρωτοβουλίες μπορούμε να λάβουμε για να βελτιώσουμε γενικά την γάμα των εργαλείων που έχουμε κοιτάμε την αμερικανική εμπειρία, ας πούμε, και την αυστραλέζικη εμπειρία, ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, διατηρήσουμε τη γεωργία μέσα στα πλαίσια αυτής της μεταβλητότητας της αγοράς. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση όσο το δυνατόν. Το περασμένο φθινόπωρο, λοιπόν, ε, δώσαμε ένα πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ ε, και είναι απογοητευτικό που δεν το χρησιμοποίησαν όλες οι χώρες ε, είναι 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε λοιπόν μία αντίδραση σε επίπεδο Ευρώπης, κανείς δεν τη χρησιμοποιεί και είναι 100% ε, χρηματοδότηση. Δεν θέλουμε να επανεθνικοποιήσουμε την ΚΑΠ, ε, είναι πάνω από τα ε, προσδοκίες τα χρήματα που δίνονται και δεν χρησιμοποιούνται. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου ελπίζω ότι τα μέλη ε, κράτη-μέλη που έχουν μισή μηδενική απορρόφηση να το κάνουν, γιατί δεν είναι προς το όφελος των αγροτών. Κάποιοι επίσης ε, χρησιμοποιούν τα χρήματα για αναδιάρθρωση του τομέα. Όμως καλύτερα να τα δώσουν στους γεωργούς, γιατί αυτοί τα χρειάζονται. Η ανισορροπία στην αλυσίδα διατροφής επίσης. Ε, ξέρετε τις απόψεις μου, τις έχω πει πάρα πολλές φορές, έχετε κάνει πολλή δουλειά στην Επιτροπή σας γι' αυτό. Και προφανώς στην Ολομέλεια θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να πούμε ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τη διατροφική ε, αλυσίδα και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και περιβάλλοντος ε, θα συζητηθεί το θέμα και περιμένω με αδειμονία αυτό το αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να έχουμε την αντίστοιχη υποστήριξη για τα μέτρα στην διατροφική αλυσίδα. Για άλλη μια φορά να πω ότι είναι μια μελέτη που κάνουμε με την Task Force, μαθαίνουμε από την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Λιθουανίας, ε, από χώρε δηλαδή που έχουν εφαρμόσει αυτά τα μέτρα για να αξιολογήσουμε. Αντίστοιχα, τώρα, για την κρίση στον τομέα των, της γαλακτοπαραγωγής. Ε, έχουμε 23 μέτρα το Σεπτέμβρη και το Μάρτιο συγκεκριμένα ήταν τελευταία φορά. Οι 100 προτάσεις που έκαναν τα κράτη-μέλη και εσείς εξετάστηκαν και είναι 23 αυτές που εφαρμόσαμε διότι οι υπόλοιπε ήταν εκτός του προϋπολογισμού και των νομοθετικών περιορισμών που έχουμε. Όμως ε, χρησιμοποίησαμε όλα τα νομοθετικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εξορρόπηση μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Και υπάρχει μια μεικτή αντίδραση, για να είμαι ειλικρινή, σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων για την εθελούσια. Και συμφωνώ ότι ο καθένας πρέπει να κάνει το δικό του, ε, να παίξει το δικό του ρόλο. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους ε, παραγωγούς για να σταματήσουν την παραγωγή, να την παγώσουν. Όμως, ο αγρότης, ο, παραγωγός θα αποφασίσει τελικά και όχι η Κομισιόν και το 85% της παραγωγής του γάλακτος καλύπτεται από αυτό το σχέδιο. Είναι αυτά που αναφέρει και ο κύριος Ντές για την Γερμανία. Τώρα, σε σχέση με το ε, διορισμούς, με, το ANC, ε, όντως, κύριε Νίκολσον, Είμαστε σε επαφή με τη Βόρεια Ιρλανδία για αυτό το θέμα. Μου το ανέφεραν το θέμα στην Βόρεια Ιρλανδία πρόσφατα, ε, το τι περνάνε δηλαδή και την περιχαράκωση αυτής της περιοχής. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ανησυχούσαν σε σχέση με τα όρια, οπότε συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Αυτά πρέπει να κάνουν προτάσεις στις περιφέρειες, αλλά η Κομισιόν πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι αρχές. Η χαρτογράφηση θα μας βοηθήσει, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε ε, πάρα πολύ στο θέμα του καθορισμού των ορίων ε, των ε, χωραφιών, για παράδειγμα. Θα αφήσουμε αυτές τις πολιτικές στην Βόρεια Ιρλανδία και τις αρχές της. Επίσης θα κάνουμε και μία συμφωνία των συσσωρευμένων επιπτώσεων ε, που θα είναι διαθέσιμη στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα έχουμε μια ιδέα σε γενικές γραμμές για το τι έχει εξεταστεί, τι έχουμε κερδίσει από τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ως τώρα και θα έχουμε ε, και μια ιδέα για το τι μπορούμε να κάνουμε στις στα μελλοντικά deal. Οι διαπραγματεύσεις TTIP, η εντολή είναι ξεκάθαρη και είναι γνωστή. Θα διατηρήσουμε τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο αξίας των ζώων, διαστροφικής ασφάλειας, βιώσιμης γεωργίας. Ε, πολλές φορές ε, δεν εκτιμάται, αλλά συνεχίζουμε να το λέμε. Είναι η αλήθεια και είναι μέλος της εντολής. Δεύτερον, να πω ότι είναι σχετικά αργές οι διαπραγματεύσεις, διότι η θέλουν να έχουν μία ε, συμφωνία πρόσβαση στην αγορά μόνο και σε όλα τα επίπεδα. Δεν τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα όπως ε, ε, το καθεστώς ενίσχυσης τα υγειονομικά ζητήματα, συγγνώμη, και όλα τα άλλα ζητήματα που αφορούν σε εμά και στο γάλα μας, γιατί αυτοί έχουν άλλα προϊόντα, τα προβλήματα που έχουμε γεωγραφικές ενδείξεις. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό και όλοι εδώ έχουν την ευκαιρία να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με το τελικό αποτέλεσμα. Το κοινοβούλιο είναι που θα αποφασίσει και το λέει και στον κύριο Χόισλινγκ. Τα 28 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, έχουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν ε, όλα αυτά. Και είναι η μόνη δημοκρατική απόφαση που μπορείτε να πάρετε και να το κάνετε αν δεν συμφωνείτε με, τη, με τον deal. Φυσικά, και η Υπουργή για το Εμπόριο πρέπει να διασφαλίσει ότι θα έχουμε τις βέλτιστες πιθανότητες επιτυχίας, ενώ θα έχουμε χάσει και σπαταλήσει χρόνο. Τώρα για την αλλαγή κλίματος στις διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα στο Παρίσι ε, δόθηκε μεγάλη όθηση για το θέμα των ε, αερίων του θερμοκηπίου και συμφωνώ ότι όντως η Γεωργία πρέπει να έχει ένα ρόλο και ότι πρέπει αυτό να γίνει με, ίσους, με όρους. Ε, να πω καταρχάς ότι συζητούμε και διαπραγματευόμαστε το LULUCF. Επίσης θέλουμε να υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, στην ε, Κομισιόν σύντομα για να, και να ληφθούν υπόψη διάφορα κριτήρια ε, για το ακασταθάριστο ε, εθνικό προϊόν και άλλα τέτοια ζητήματα που θα συνεισφέρουν ε, στη συζήτηση, τα οποία είναι πολιτικά, αλλά όμως υπάρχουν και συγκεκριμένοι επιστημονικοί λόγοι που καθορίζουν πώς όλα αυτά θα συντεθούν. Όμως δεν μπορώ τώρα να σας πω περισσότερα γιατί δεν έχουν βγει συμπεράσματα. Όμως σημειώνω το γεγονός ότι πρέπει πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια και δικαιοσύνη. Για την ε, επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και το ερώτημα που θέσατε, δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δώσαμε ευελιξία στην τελευταία μεταρρύθμιση και μεγάλο βαθμό επικουρικότητας, διότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία μέσα από τις διαπραγματεύσεις αν δεν υπήρχε αυτό. Αν είχαμε μία ΚΑΠ που θα ήταν για όλους η ίδια, ε, δεν θα υπήρχε συμφωνία. Οι πιο ισχυρές ε, βέβαια ε, οικονομίες ε, ε, υπερισχύουν των ασθενών οικονομιών γιατί έχουν πολλά χρήματα στον κορβανά τους και σε επίπεδο χρηματικών πόρων, δεν θα δώσω ονόματα χωρών, αλλά κάποιες χώρες είναι πιο ισχυρές από άλλες. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια ε, απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά καιρού και αυτό έκανα πέρυσι το Σεπτέμβρη. Έδωσα λοιπόν κάποιου πόρου με βάση κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη αυτό το πράγμα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν όμω με τον τρόπο που έπρεπε. Και ε, αν δεν δαπανηθούν τα χρήματα του Σεπτεμβρίου δεν ξέρω αν θα ξαναπάρουμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Συμφωνώ ότι δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε μια πλήρη επανεθνικοποίηση των αντιδράσεων στα γεωργικά προβλήματα, γιατί ε, θέλουμε να έχουμε ίσους όρους ε, για όλους τους πολίτες ε, στην Ευρώπη, όχι μόνο τους γεωργούς, γιατί η γεωργική πολιτική είναι ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Δεν καταλήξαμε ακόμη σε συμπέρασμα για το τι θα πρέπει να έχει αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση. Πάντως θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια εργαλεία διαχείρισης των κρίσεων, να βοηθήσουμε τους γεωργούς της επιχειρήσεις ε, για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να ανταποκριθούν πιο γρήγορα στα προβλήματα της αγοράς που αντιμετωπίζουμε σε πολλούς τομείς. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της απλούστευσης και να μειώσουμε την περιπλοκότητα των πολιτικών μας, ε, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητά τους ε, και ιδιαίτερα την περιβαλλοντική τους αποτελεσματικότητα. Και θα πρέπει να γνωρούμε το γεγονός ότι οι διεθνείς συμφωνίες, ε, είχαμε το 2015 πολλά θέματα για τους βιώσιμους στόχους της χιλιετίας, για τις κλιματικές αλλαγές, θα πρέπει να λάβουμε και εμείς ενεργό μέρος στην εφαρμογή αυτών των συμφωνιών που έχουν συναυθεί. Και θα καθορίσουν και αυτές τις τι μελλοντικέ κατευθύνσεις των πολιτικών μας. Κυρία Σένρα Ροντρίγκε, αν έχετε αποδείξει για παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού στην Ισπανία, ιδιαίτερα στη Γαλλικία, παρακαλώ μεταβάστε στις ε, ε, ευρωπαϊκές αρχές ε, και καλό θα ήταν οι αρμόδιοι να διερευνήσουν τις υποθέσεις αν όντως υπάρχουν στοιχεία και δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε για αδικοπραξίες. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές βοήου και μοσχαρίσιο κρέατος, όντως ε, υπάρχει πρόβλημα και ακριβώς αυτή η μελέτη σωρευτικών επιπτώσεων που θα κάνουμε για τις συμφωνίες ελευθέρω εμπορίου θα καλύπτουν όλα τα προϊόντα και φυσικά και το βόιο. Μάλιστα στο πλαίσιο της συμφωνίας Μερκοσούρ αφαιρέσαμε το βόλιο γιατί μειώνεται η ζήτηση βοηθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητούμε αύξηση των εισαγωγών βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισορροπία μεταξύ τη παραγωγή βοηθού κρέατο, τη κατανάλωση και των εισαγωγών βοήου κρέατο. Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η σχετική έκθεση. Ελπίζω να απάντησε σε όλε τι ερωτήσει, κύριε Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, για τη Ρωσία, για το ρωσικό εμπάργκο. Εγώ δεν αποποιήθηκα των ευθυνών μου. Γνωρίζω ποιο είναι υπεύθυνο και αρμόδιος και γιατί. Ο κύριος Ανδριοκάητης, ο Επίτροπος Ανδριοκάητης συναντήθηκε πρόσφατα στο Παρίσι με τον, ε, Επίτροπο, ε, με τον Υπουργό Γεωργία της Ρωσίας ε, σε μια διάσκεψη. Πρόοδο δεν υπήρχε, αλλά αυτό δεν οφείλεται στον κύριο Ανδριοκάητες, στον Επίτροπο Ανδριοκάητες. Πολλές συνομιλίες γίνονται, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν έχουν δεσμευτεί ακόμη για να εξομαλύνουν τις εμπορικές μας σχέσεις ε, και να τις ανάγουμε στο, στο επίπεδο του παρελθόντος. Τώρα, για τα αυγά δεν είμαι ειδικό, θα το κοιτάξω. Πάντως είναι περισσότερο θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας, ε, Σάντε. Αν πάντως έχετε λεπτομέρειες για τεχνικά θέματα, για το χρώμα του και πολύ ευχαρίστως να τις διαβιβάσω στον Επίτροπο Ανδρουκάητες για να σας απαντήσει. Εγώ στηρίζομαι σε επιστημονικά πορίσματα για τη γλυφοσάτη και, για αυτό το θέμα αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον αν μονομερός η Γαλλία αποφασίσει να απαγορεύσει εισαγωγή προϊόντων που έχουν στα οποία χρησιμοποιηθεί η γλυφοσάτη και στο παρελθόν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο με άλλα φυτοφάρμακα. Και η Υπουργό Σεγκολέν Ροϊάλ απαγόρευσε την εισαγωγή αρκετών προϊόντων. Πάντως δεν έχουμε ακόμη καταλήξει το θέμα αυτό. Ακόμη περιμένουμε διευκρινήσεις από μερικά κρατημέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συγκεκριμένων επιστημονικών προϊόντων και του συγκεκριμένου προϊόντος. Και δεν ξέρω αν θα σκόπιμο ε, αυτό το προϊόν να εγκριθεί και πάλι για χρήση. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ένα λεπτό καθένας παρακαλώ. Αποφύγετε τις επαναλήψεις για να κερδίσουμε χρόνο. Η κυρία Εράνς Γκαρσία, ένα λεπτό επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε. Ε, σε χαλεπούς ε, καιρούς αναλάβατε τα καθήκοντά σας ε, για τη γεωργική πολιτική. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σε σχέση με μία φήμη που ακούγεται για το μέλλον της ΚΑΠ και της, του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Τι γίνεται, η αγροτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη πέτρου θα περάσει την περιφερειακή πολιτική και θα περάσει και το ε, το γεωργικό εμπόριο στην διεύθυνση εμπορικής πολιτικής. Τι θα γίνει με τη Γεωργία. Για το τι έχουμε προχωρήσει καθόλου στις γεωγραφικές ενδείξεις. Μάλλον όχι. Άρα δεν, έχουμε πάρει στραβό δρόμο. Αν θέλουμε ε, συμφωνία μέχρι τα τέλη του χρόνου θα πρέπει να πιέσουμε πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς. Σε ό,τι αφορά το γάλα, ε, α, οι επιχειρήσεις μας απειλούν με έξοδο από την Ισπανία και με την κατάσταση. Τι θα γίνει ε, σε ό,τι αφορά το παρατηρητήριο των τιμών. Ζητήσαμε με έκθεσή μας ε, τη σύσταση παρατηρητηρίου των τιμών. Θα ήταν πολύ χρήσιμο. Τι γίνεται. Επίση, μιλήσατε για ανάψματα σε παραγωγού. Τι εννοείτε. Θα δοθούν νέα κονδύλια πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ για να προωθηθεί η μείωση της παραγωγής. Είναι φρέσκα να πω χρήμα, γιατί μόνο έτσι θα δώσουμε κίνητρα στους γεωργούς για να μειώσουν την παραγωγή τους. Και τέλος, με τέτοιες τιμές παρέμβαση σε απορροκυπευτικά και γάλα δεν, πρόκειται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση των τιμών. Ευχαριστώ. Κυρία Σράερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας βλέπω σήμερα. Μιλάμε για την κρίση στη Γεωργία. Μιλάμε για τον γαλακτοπαραγωγικό τομέα. Στην πραγματικότητα μιλάμε για κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Πολλοί θέλουν να σταματήσουν να ασχολούνται με τη γεωργία και δεν τα καταφέρνουν. Καθημερινά φτάνουν στα αυτιά μας τέτοιες ιστορίες. Ιστορίες οικογενειακές που είναι δυσάρεστες. Δεν θα ήταν καλύτερα να πάρουμε τα χρήματα, ε, τα επιπλέον για την υποστήριξη που προβλέπονται και να τα χρησιμοποιήσουμε στην κοινωνική και οικονομική μας πολιτική. Ας βοηθήσουμε τους Γιώργους να πάυσουν τις δραστηριότητε τους και να ασχοληθούν με κάτι άλλο για να υπάρξει και καλύτερη ισορροπία στην αγορά. Κοιτάξτε τι γίνεται με το γάλα, με το χείριο. Περισσότερη ισορροπία χρειαζόμαστε. Αυτό το έχουν υποστηρίξει πολλές διαφορετικές πηγές. Μιλήσατε και για τη Ρωσία, είπατε. Ότι φταίει ο Ρώσος υπουργό. Όμω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πιστοποιητικά εξαγωγικά από τα ίδια τα κρατημέλη. Δεν θα μπορούσαν τα κρατημέλη να έχουν δημερό συμφωνίε με τη Ρωσία. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειαζόταν να περνάμε όλο αυτό το, ε, όλη αυτή τη διαδικασία και το λαβύρινθο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν πιο εύκολο να βελτιώσουμε την κατάσταση έτσι, διμερό. külső állomásain. Itt vagyok biztos úr, tisztelettel a másik oldal. σας ε, ε, επιστήσω την προσοχή. Εδώ κάθομαι, σε αυτή την πλευρά, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έγιναν κάποιες δοκιμές και σύμφωνα με αυτές τις δοκιμές ε, διαπιστώθηκε ότι το 31% του μελιού είναι νοθευμένο. Αυτό ε, δόθηκε ως στοιχείο στις 11 Μαΐου. Κάθε ε, χρόνο μπαίνουν 165.000 κιλά ε, θευμένου ε, μελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μια τέτοια ε, ποσότητα όταν πωλείται στην εσωτερική αγορά θα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ άσχημο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα και σε σχέση με την Γαλλία. Ο κύριος Μπέλντερ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Φαίνεται ότι ξεκινήσατε μια διπλωματική προσπάθεια για να αυξήσετε τις ε, εξαγωγές μας προς την Κολομβία, την Κίνα, την Ιαπωνία και μάλιστα θα πάτε και στην Ινδονησία και το Βιετνάμ. Μέχρι στιγμής είχαμε τα αποτελέσματα. Είστε ικανοποιημένος από αυτές τις διπλωματικές σας προσπάθειες και ποια θα είναι η εμπορική σας πολιτική για το 2017. Η κυρία Ντότς. Η κυρία Ντότς. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Στη Βόρεια Ιρλανδία, στην εκλογική μου περιφέρεια, πρόσφατα είχατε έρθει για να μιλήσετε για το Brexit. Αν είχατε μείνει λίγο παραπάνω, όπως και εγώ, θα παρακολουθήσετε και το γεωργικό, τη γεωργική έκθεση που έγινε στο Όλστερ και θα είχα την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή και με γεωργούς. Εκεί θα ακούσετε τον ένα γεωργό μετά τον άλλο να μιλούν για τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν κυρίως εξαιτία των χαμηλών τιμών, της αστάθειας των τιμών και της έλλειψης ρευστού. Και αισθάνονται ανήμποροι και καταλελειμμένοι. Και πολύ απογοητεύτηκα από τα σημερινά σας σχόλια. Σε ό,τι αφορά την, ε, την οικειοθελή ε, συμμετοχή στη διαχείριση, πιστεύετε ότι χωρίς στρατηγική καθοδήγηση από το Συμβούλιο δεν θα, θα είναι αρκετό με ένα εκούσιο σύστημα να βρούμε λύσεις. Και σε ό,τι αφορά την διάμεση αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής, Σίγουρα χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο δραστικό από κάποιες μικροπροτάσεις που υποβάλλατε σήμερα. Ευχαριστώ, η κυρία Πετήρ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Από τον Απρίλιο, μέχρι τον Απρίλιο μάλλον, είχαμε συνεχείς παγετούς στην Ευρώπη ε, και πολλές πλημμύρες και άλλα αρνητικά καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα σας ενημέρωσα για το πρόβλημα του παγετού που είχαμε και για τις ζημίες ε, στην Κροατία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, την ε, Ρουμανία και την Ουγγαρία. 800 περίπου εκατομμύρια ήταν οι ζημιές, μέχρι και ένα δισεκατομμύριο υπολογίζουν μερικοί. Επιλήγησαν κυρίως οι αμπελουργοί μας και επιπλέον αυτά προστίθενται στη, στο ρωσικό εμπάργο και στην και στην αστάθεια των τιμών και στα προβλήματα της αγοράς και αυτές οι κακοκαιρίες ε, και οι θεομηνίες πραγματικά γονάτισαν τους γεωργούς μας. Έχουν ε, υποβληθεί πολλές αιτήσει για βοήθεια. Πώς ε, θα βοηθήσετε τους γεωργούς μας που έχουν πληγεί επιπλέον και από τους παγετούς και τα χαλάζια, γιατί δημιουργήθηκε περαιτέρω διαταραχή των αγορών εξαιτίας αυτών των θεομηνιών. Πιστεύετε ότι μπορούν να ληφθούν όλα αυτά υπόψη στο γεωρικό προπολογισμό και μάλιστα να αναζητηθούν νέε πηγέ χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντενανό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μα σε μια περίοδο τόσο παραγμένη. Να μην τι άλλο για τη Γεωργία. Η κατάργηση των γαλακτοπαραγωγικών ποσοστώσεων έχει ήδη δείξει τι συνέπίε τη περισσότερη παραγωγή, αλλά μείωση των τιμών. Να μην έχουμε αυταπάτες. Χρησιμοποίησατε το άρθρο 222 των ενιών ΚΟΑ, αλλά δεν εξαρκεί σήμερα. Πρέπει να αναζητήσουμε απαντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλλον πρέπει να βοηθήσουμε με, κοινοτικές, με κοινοτικά κονδύλια, όσα διαθέτουμε, την Γεωργία δεν πρέπει να επανεθνικοποιηθούν οι γεωργικές πολιτικές. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι αντικείμενο ε, προστασίας. Έτσι θέλω να το δείτε, να την προσπιστείτε και από την πλευρά του προπολογισμού. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Προπολογισμών και ξέρω τι σας λέω. Η ε, δέσμευση πιστώσεων εδώ ή εκεί και η μετακίνησή τους μπορεί να οδηγήσει στη χρηματοδότηση άλλων πολιτικών. Θα πρέπει λοιπόν να ε, σκεφτείτε και το άλλο. Μήπω αναγκάζετε του ε, γεωργού να πάνε πολυτεχνείο για να μπορούν να συμπληρώσουν τη δήλωσή του για τι βοηθείες τη ΚΑΠ. Ο κ. Φεράν, ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Μερικέ σκέψει γιατί άκουσα ένα συνάδελφο να λέει ότι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και λιγότερη δημοκρατία. Εγώ έχω διάθεση να το απαντήσω. Όσο περισσότερη Ευρώπη υπάρχει, τόσο περισσότερο λιγοστεύει η δημοκρατία. Κύριε Επίτροπε, Πρέπει να αναφερθώ σε κάποιες από τις δηλώσεις σας. Μιλήσαμε για μια ε, προσέγγιση ενιαία. Τα κράτη-μέλη έχουν αναθέσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπραγματευτούν ε, εμπορικέ συμφωνίε που όμω έχουν τελείω αντικρούμενα συμφέροντα για τι εισάγουσε χώρε και για του παραγωγού. Θα πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι, λέτε, και να παραμείνουμε φιλόδοξοι κυρίω στην ουσία και όχι στο ρυθμό. Μετά την παρέμβασή σα όμω, κύριε Επίτροπε, δεν καταλαβαίνω γιατί το μοντέλο των ελεγχόμενων γεωγραφικών αντίξεων που είναι καθοριστική σημασία για μα και που ισχύει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αμφισβητηθεί. Ε, ωστόσο, Επίτροπε, οι διπλωματεύσεις των Συμφωνίας τύπου που συνεχίζονται από διαφορετικέ πηγέ επιβεβαιώνουν ότι οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σε αυτό το ζήτημα και ότι το θέμα δεν έχει καν αρχίσει να θίγεται. Είτε είστε μάγος και ταχυδακτηλουργός, είτε δεν μας λέτε την αλήθεια. Έχω δύο ερωτήσει λοιπόν, Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα, οι ενδείξεις, οι ονομασίε αυτέ που είναι το ε, αναπόσπαστο κληροδότημα της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να συζητιώνται στις διαπραγματεύσει. Και δεύτερη ερώτηση, γιατί μόνο με αφορμή αυτές τις διαπραγματεύσει έχει ε, δημιουργηθεί ένας κατάλογος κλειστός και όχι ένας κατάλογος που να καλύπτει όλες τις υπάρχουσες γεωγραφικές ενδείξεις. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χόιμπουχ. Η κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να θίξω τώρα ένα άλλο διαφορετικό θέμα, την συγκέντρωση της γης και την αρπαγή της γης. Η Επιτροπή Ε, επέκρινε την μελέτη της ε, Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου ότι δεν υπήρχε μία βάση με δεδομένα και θα ήθελα να διαφωτίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, Εν ώψη του γεγονότος ότι έχουμε πολύ λίγα δεδομένα και μια μικρή βάση ε, υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα και επαρκή ε, δεδομένα. Ε, πότε θα μας τα διαθέσετε, πότε θα αρχίσετε να τα συλλέγετε σχετικά με, το να, με τις συναλλαγές, ποιοι είναι οι αγοραστές, πόσα εκτάρια, ποιος είναι αυτός που πουλάει και ποιες είναι οι τιμές ε, για τη γη που δίνονται, ε, το θέμα της διαφάνειας, ε, της λήψης γης, της συγκέντρωσης γης, γιατί η γη είναι η βάση για τη γεωργία και το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ που ήρθατε για ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Έχω σχόλιο και μια ερώτηση. Στον, ε, στο άρθρο 32 του κανονισμού ΠΟΖΕΙ προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αναλύσει ιδιαίτερως τα θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές με βάση ε, μελέτες που θα αποτελέσουν βάση για την προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες εμπορικές διαπραγματεύσεις. Με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμ, εμφαρμόζει αυτή αυτό το άρθρο στα πλαίσια των συμφωνιών και των διαπραγματεύσεων Μερκοσούρ και TTIP, γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Και το σχόλιο μου αφορά τις τιμές του γάλακτος που έχουν φτάσει ιστορικά να αναδύρ η κατάσταση είναι ανυπόφορη για του κολακτοπαραγωγού. Τα κράτη-μέλη καταβάλουν ε, χρηματοοικονομικέ προσπάθειες, το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν αρκεί αυτό για να αναχαιτιστεί η περαιτέρω μείωση των τιμών και να αμείβονται δίκαια για την εργασία του οι γεωργοί μα και οι κτηνοτρόφοι μας. Κύριε Επίτροπε, ε, πιστεύω ότι μετά την ε, κατάργηση των ποσοστώσεων το, το σύστημά μα δεν λειτουργεί σωστά η αυτορύθμιση δυστυχώς ε, έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλμένη. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Δαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Η παρούσα κρίση ε, καταδεικνύει για μία ακόμη φορά τις ε, ε, τα προβλήματα υπάρχουν σχέση μεταξύ παραγωγών και αγοραστών. Από την συνθήκη της Ρώμης είχαμε προβλέψει συγκεκριμένες διατάξεις ε, στο δίκαιο του ανταγωνισμού για να επιτρέψουμε τους, τους ε, γεωργούς μας να οργανωθούν και να διαπραγματεύονται πίσω όρις με τους αγοραστές τους. Διαπιστώνουμε όμως ότι αυτή η ιδεώδης κατάσταση ανήκει στη φαντασία μόνο. Στην τελευταία μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε αυτές τις ε, διατάξεις για τις οργανώσεις ε, των παραγωγών και να βελτιώσουμε ε, τις διατάξεις του δικαίου ανταγωνισμού καθιστώντα τι πιο ευνοϊκέ για τους γεωργού. Έχουμε όμω την αίσθηση ότι εξακολουθούν να υφίστανται πιέσεις η Γεωργία και να μην μπορεί να κάνει τίποτα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού που είναι ήδη υπερφορτωμένη. Πώς μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον το δίκαιο του ανταγωνισμού προς όφελος και προς εξυπηρέτηση των γεωργών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω άλλη μια φορά για την TTIP, την ε, Συμφωνία Ελευθέρου ε, εμπορίου. Πάρα πολλές φορές μιλήσαμε για τις γεωγραφικές ενδείξεις σήμερα και στις συμβάσεις ε, που συζητούνται στις διαπραγματεύσεις για την TTIP αναφέρεται το θέμα της προέλευσης, όμως ε, είναι μεγάλο μυστικό πώς ε, τελικά δημιουργήθηκε αυτή η λίστα. Η λίστα και στις δύο ε, συμφωνίες στην ουσία δεν μας δείχνει ποια είναι η προέλευση των προϊόντων που πηγαίνουν ας πούμε στην Καναδά, στην Νότια Αμερική, στο Βιετνάμ. Θα μπορούσαν να είναι λοιπόν μία λίστα ε, η οποία θα είχε αυτά τα στοιχεία για να μπορεί να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς. Ε, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η λίστα και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε για να ε, αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάζεκαμπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε και άλλες γεωργικές κρίσεις και σε άλλους τομείς. Έχουμε την κρίση με το πόσιμο είδωρο, έχουμε την περιβαλλοντική κρίση και αν λάβω τις κατοχώρες ως σημείο αναφοράς, βλέπω ότι πόρο έχουμε ακόμη από την τήρηση των διεθνών μας δεσμεύσεων και συμφωνιών. Και θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Στην οδηγία πλαίσιο για το νερό και στην οδηγία για την ε, ποιότητα του αέρα. Η, η εντατική κτηνοτροφία ρηπαίνει ιδιαίτερα και το νερό και το περιβάλλον. Και μάλιστα αν ενισχύσουμε την ε, παραγωγή στην κτηνοτροφία σίγουρα θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ανοιχετήσουμε αυτήν την υπερπαραγωγή. Επίσης, ε, αν συνεχιστεί η παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης, τότε θα πρέπει να, χαιρετήσουμε, να αποχαιρετήσουμε την βιοπικιλομορφία μας. Το μέλλον της είναι μαύρο ζωφερό παρά πράσινο. Φαντάζομαι ότι προτιμάτε το πράσινο από το μαύρο. Ο κύριος Στάκουλα. Joo, kiitoksia <clears throat> komissaarille hyvästä kattavasta tilannekatsauksesta ja Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ε, συνολική επισκόπηση. Ευχαριστώ για τις ε, δράσεις που έχετε αναλάβει, κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση στην αγορά των ε, γαλακτοκομικών και του χείρου κρέατος είναι σοβαρή, για να μην πω Η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει αν σε τοπικό επίπεδο γινόταν υψηλότερες πληρωμές στους παραγωγές, ας πούμε, στο, το 2016. Οι προστοβαρείς ε, ε, πληρωμές είναι μια επιλογή η Φιλανδία το ζήτησε αυτό πέρυσι και θα έπρεπε να μπορεί να το κάνει και φέτος. Είναι προκαταβολές στην ουσία, όμως ε, απαιτούν αλλαγές στο σύστημα μηχανογράφησης. Πέρυσι έγιναν πολύ αργά και λίγοι ήταν οι γεωργοί που τα κατάφεραν. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να κάνει μια μελέτη σχετικά με την εμπροστοβαρής ε, πληρωμές. Κύριε Χόγκαν, είστε έτοιμος για κάτι τέτοιο. E, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε και στη Λιθουανία, συναντήσατε Λιθουανούς γεωργούς και συζητήσατε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα σήμερα το πιο δυνηρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το εξής. Η γαλακτοπαραγωγή και οι γεωργοί μα έχουν χάσει την ανταγωνιστικότητά του εξαιτία τη μείωση των τιμών. Οι τιμέ βρίσκονται στον ΑΔΙΡ και οι πληρωμές, ενισχύσει είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ε, ε, οδηγείται σε εξαφάνιση ο γαλακτοκομικός κλάδος στη Λιθουανία δυστυχώς. Τι μπορούν να περιμένουν να η γεωργική γαλακτοπαραγωγή της Λιθουανίας θα αυξηθούν επιτέλους οι τιμές, γιατί οι διαφορές ε, στις τιμές μεταξύ βαρτικών χωρών και υπόλοιπων χωρών είναι μεγάλες. Και μάλιστα η λιθουανική γεωργία έχει χάσει απόλυτα την ανταγωνιστικότητά της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ε, Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω ε, να πω εξ αρχής ότι το να είσαι ριζοσπαστικός δεν είναι ένα καλό μέσο. Ε, δεν χρειαζόμαστε μία ριζοσπαστική ε, αναστροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική χρειαζόμαστε τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε να τα επεξεργαστούμε και να έχουμε συγκεκριμένα ε, βήματα που θα κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Χαίρομαι για την απλούστευση για τη δυνατότητα να δίνονται ενισχύσεις μέσα από τα κράτη-μέλη, όμως δεν θεωρώ ότι ε, φτάνει ε, αυτή η δυνατότητα μέσα σε 6 με 12 μήνες να δίνεται. Πρέπει να το επεκτείνουμε αυτό. Αν ε, λοιπόν θεωρείτε κι εσείς ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τον κανόνα de minimis, να τον διπλασιάσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την υπαρξιακή κρίση της γεωργίας. Ευχαριστώ κύριε Σκαλινόφσκι. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, Πιστεύω ότι η εξάλληψη των γαλακτοκομικών ε, ε, ποσοστώσεων σε συνδυασμό με το ρωσικό εμπάργο ε, οδήγησε σε αυτή την τεράστια κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα. Με θύματα τους γεωργού μας φυσικά. Ε, ερωτώ, συμμερίζετε τους φόβους των παραγωγών ζαχαροτεύ, ε, ε, παντζαριών, ζαχαροτεύτλων μάλλον στην Πολωνία γιατί φαίνεται ότι οι παραγωγές αλλάζουν από τη μία χώρα στην άλλη, ε, όχι λόγω ανταγωνιστικότητας, αλλά λόγω ιδιοκτησίας ε, του κεφαλαίου. Και αυτό φέρει σε δύσκολη θέση τους ε, παραγωγούς συγκεκριμένων χωρών. Επίσης, από τη μία καταργούμε τις ποσοστώσεις μας και από την άλλη ανοίγουμε διαπραγματεύσεις ελεύθερο εμπορίο. Αυτά δεν πιστεύετε ότι έρχονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο το οποίο μας είναι τόσο προσφυλές και προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε γιατί είναι δύνατο να τα καταφέρουμε με, τέτοιο, με τόσο αντιφατικές συμπεριφορές. Σας ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν ε, δυσκολίε με τη συμπλήρωση των εντύπων από του γεωργού. Ε, Δυστυχώ εκτό μικροφώνου ο, ε, ο μιλητή. Εκτό μικροφώνου. Στη Ρουμανία απαγορεύτηκαν οι ενισχύσει του πρώτου πυλώνα ε, λόγω τη δυσκολία υποβολή των εντύπων. Έχουν ακόμα 200.000 αιτήσει πληρωμών που δεν έχουν πληρωθεί στου γεωργού. Και αυτό ισχύει και για τα ζωοτεχνικά και για την ίδια τη γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω τις εξής ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα αιτήματα των ρωμανικών αρχών και διαθέτεται και μηχανισμό για να διορθώσετε αυτή την κατάσταση. Όμως, για τα πλήρωτα, για τα μη καταβληθέντα ποσά, για αυτά τα εκατομμύρια ευρώ, πώς και δεν έχει καταβληθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ από όλα αυτά τα ποσά. Ο κύριος Φλάναγκαν, ευχαριστώ πολύ. Επίτροπη, Επιτροπή, καλό είναι να κάνει θετικό, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να είναι ρεαλιστή. Τον Ιανουάριο του 2015 μα είπατε ότι δεν υπάρχει κρίση στο χαρακτοπραγικό τομέα. Τώρα μα τα λέτε αλλιώ. Και αλλάξετε γνώμη. Παραδεχτήκατε ότι υπάρχει κρίση στην Γεωργία φέτο, μέσα στη χρονιά. Και λέτε τώρα να είμαστε θετικοί, γιατί οι εξαγωγέ ε, για τα διάφορα γαλακτοκομικά ε, αυξάνονται. Τι νόημα έχει αυτό, εάν οι παραγωγοί ε, παράγουν και δεν βγάζουν τίποτα, διότι χάνουν χρήματα. Και πώ να είμαστε θετικοί για αυτό το πρόβλημα, όταν κάποιοι πολλούν τα προϊόντα του τελικώ με χαμηλότερο κόστο και δεν λύνουν το πρόβλημά του. Για μένα αυτό είναι η ουσία του θέματο. Και για την απλούστευση μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι έχουμε διαρθωμένο διάλογο, οπότε θα ήταν καλό να ξαναδούμε τα αγγλικά που φαίνεται ότι οι λέξεις της παραποιούνται. Γιατί δεν κοιτάτε να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ε, ένα μεγαλύτερο ποσοστό σφάλματος ε, στις διάφορες μετρήσεις. Με το Brexit επίσης, τι θα γίνει εφόσον συμβεί και πώς θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες. Και όπως ε, μιλάτε εσείς για το εθνικό σας κράτος, εγώ είμαι εδώ εκπροσωπώντας στην Ιρλανδία όσο και εσείς στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστώ. Κυρία Μίλλερ, κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το μαθητικό πλώσιο και χρησιμοποίησατε όλα τα εργαλεία στη χρηματοδότηση. Είπατε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα ε, στον προπολογισμό εκτός από αυτά τα 420 εκατομμύρια Μύρια ε, ευρώ μιλήσατε για τις συνδεδεμένες πληρωμές ε, ε, για τα κράτη-μέλη, όμως όταν κοιτάμε χώρες όπως η Φιλανδία και η Πολωνία μονομερός που δεν έχουν δοθεί ε, αυτά τα 420 εκατομμύρια καταναβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Για τη Μερκοσούρ και την TTIP ε, να πω ότι υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις όπως είπαμε ίσως να έπρεπε να έχουμε και με την Ουκρανία και άλλες τέτοιες χώρες ε, για να μπορέσουμε ε, να δούμε επίσης τι μπορούμε να δώσουμε ως κίνητρα για τις εκτάσεις που δεν έχουν κάποιον διάδοχο, επίσης ε, για, τις υποχρεωτικές, ε, για τα υποχρεωτικά όρια ποσοτήτων ήρθε καιρός να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί αν υπάρχει ε, μείωση των ε, ποσοστών στο γάλα. Ε, κυρία Ποσελάη, ευχαριστώ κύριε Πύρμη. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, ε, επισημάσεις. Είπατε ότι υπάρχουν 8 κράτη-μέλη που δεν πήραν τα χρήματα που έχετε θέσει διαθέσιμα. Υπάρχει απάντηση στην ερώτηση. Θεωρείτε ότι τα κριτήρια πρόσβασης δεν είναι αρκετά ελκυστικά, ίσως να είναι και αποτρεπτικά για κάποια κράτη-μέλη. Μια άλλη παρατήρηση σχετικά με τον γαλακτοκομικό τομέα. Να για την ανάγκη να ε, συνδέσουμε την πρόσβαση στην παρέμβαση ε, με τις ποσότητες. Ο συνάλφος Μισελ Νταντάν αναφέρθηκε στον ε, ανταγωνισμό και στον δίκαιο που πρέπει να προσαρμοστεί στι ανάγκε τη αγορά. Ο συνάδελφο από την Κροατία επίσης κύριε Επίτροπε αναφέρθηκε στι ευρωπαϊκέ ε, περιοχέ, ε, ειδικά αυτέ από τι οποίε εγώ προέρχομαι την τελευταία φορά ε, είχαμε στην καλλιέργεια, το ε, πάγωμα των ε, αμπέλων που ήταν πάρα πολύ ε, πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριος Κοντζενούκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Κουσμιούκ. είπατε από την πλευρά σας ότι η Κομισιόν θα προσπαθήσει να ανοίξει η Αμερικανική αγορά για τα αχλάδια και τα μήλα στην Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά εν ώψη του ρωσικού εμπάργκο. Ε, έχουμε πρόβλημα με τις εξαγωγές σε αυτό το τομέα. Ε, κατά τη διάρκεια, τι γίνεται με αυτές τις διαπραγματεύσεις, συνεχίζουν, έχουν αναβληθεί ε, και ποιες είναι οι προτάσεις, έχετε εργαστεί επί μέτρο και υπάρχει και ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό ε, μέχρι τα τέλη του έτους δεν θα έχει εξαντληθεί. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις μέτρα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τους γεωργούς σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το έκτακτο αποθεματικό. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρτίνες, βλέπετε αυτή τη σελίδα από ένα περιοδικό της Γαλλικής ε, που είναι από τις ε, βασικές ε, περιφέρειες γαλακτοπαραγωγής στην Ευρώπη και μάλιστα στη Γαλλικία οι κτηνοτρόφοι παίρνουν τις χαμηλότερες τιμές γάλακτος σε ολόκληρη την Ισπανία. Επίσης αναγκάζονται να αφήσουν τις αγελάδες τους να πεθάνουν στην πείνα γιατί δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές. Και επιπλέον αντιμετωπίζουν και κυρώσεις και πρόστιμα εξαιτίας κακομεταχείρισης των ζώων. Ξέρετε τι λέει αυτή αυτή, τη, αυτή η αφίσα, ότι αν είναι έγκλημα να εγκαταλείπει κανείς το κοπάδι του, δεν είναι έγκλημα να εγκαταλείπει τον κτηνοτρόφο. 65 ε, ε, γεωργοί το μήνα εγκαταλείπουν τις δραστηριότητες. Ε, ο το, ο γαλακτοπαραγωγικός τομέας αντιμετωπίζει μια κρίση που τον οδηγεί σε αργό θάνατο και μάλιστα δυστυχώ δεν καταφέραμε να αναχαιτήσουμε την κρίση αυτή τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν μπορείτε να ισχυρίζετε ότι προστατεύετε και υπερασπίζεστε τους γεωργούς. Δεν μπορείτε να λέτε ότι είστε στο πλευρό των αδυνάμων με ωραία λόγια και ταυτόχρονα να βοηθάτε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της αλυσίδης ε, διανομής, να απελευθερώνετε τις ε, ε, ε, αγορές και να συνάδεται κρυπτό και παραβίστο εμπορικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και τον Καναδά δεν πιστεύετε ότι η διατροφική μας κυριαρχία, η περάσπιση των γεωργών, η στήριξη του εμπορίου ε, βραχίας αλυσίδας δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος ε, για τη γεωργία μας. Έχετε την πολιτική ευθύνη κύριε Επίτροπε να αποδείξετε και με έργα και όχι μόνο με λόγια ότι είστε έτοιμος να σώσετε από το θάνατο τη γεωργία μας και τους γεωργούς μας ξεπεράσετε το λεπτό που είχατε. Μιλήσατε για ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Ο κύριος Μέλλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χείριο κρέα, γαλακτοκομικά, ε, πολλέ δυσκολίε στην αγορά αυτή τη στιγμή, χαμηλέ τιμέ. Οι γεωργοί απαιτούν απαντήσει. Πρέπει να θυμίσω ότι στην Πορτογαλία, ιδίω στο γαλακτοκομικό τομέα, υπάρχουν ε, περιοχέ που εξαρτώνται από αυτή την παραγωγή. η Ασόρε, η περιοχή του Μίνιου, δεν είναι σειρά μου. Έχει περιοχές λοιπόν που εξαρτώνται ιδιαίτερως από όσα συμβαίνουν. Με συγχωρείτε, έβλεπα ένα νεύμα από το Προεδρείο και νόμιζα ότι είναι για μένα. Καλύτερα. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές που εξαρτώνται πολύ από τη γαλακτοπαραγωγή. Θέλω να ρωτήσω το εξής. πρέπει να προβλέψουμε μία γραμμή αποπληρωμής για τους γεωργούς για να ελαφρύνουμε το άχθος τους ή να ξαναδούμε την στήριξη, την ελάχιστη στήριξη που μπορεί να τους δοθεί ως βοήθεια. Όμως, επίτροπε, για την ανάπτυξη τη υπαίθρου που είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ε, η Πορτογαλία με την νέα κυβέρνηση έχει προβλέψει μέτρα στήριξης με κοινοτικά κονδύλια που κατά 100% χρησιμοποιούνταν ω τώρα ενώ η κυβέρνησή μα έχει λάβει διαφορετικέ αποφάσει. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, Επίτροπε, τι μπορεί να κάνει η τωρινή πορτογαλική κυβέρνηση σε σχέση με τα μέτρα που είχε λάβει η προηγούμενη για να εξασφαλίσει τη στήριξη της Πορτογαλίας στον τομέα που τώρα έχει τόσο πολύ πληγή. Ο κύριος Καπούτα, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ επίτροπε Χόγκαν για την ε, ευγενική καλοσύνη με την οποία προσέρχεστε σε αυτή την επιτροπή. Παρεμβαίνω ως ακροτελεύτιος αγορευτής, γιατί έχουν ήδη τεθεί πολλές ερωτήσεις, οπότε δεν θέλω να τις επαναλάβω. Ήθελα απλώς να εκφράσω την ανησυχία, την ανησυχία μου για τις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Πολύ συχνά μιλούμε μόνο για την συμφωνία TTIP και παραγνωρίζουμε άλλες συμφωνίες, όπως αυτή με τη Μερκοσούρ. Θεωρώ ότι για την κοινή αγροτική πολιτική είναι μία συμφωνία εξαιρετικά σημαντική. Αν σκεφτούμε το 50% των εισαγωγών από τη Μερκοσούρα έχουν να κάνουν με γεωργικά προϊόντα. Και ε, ο εμπορικό όγκο αγγίζει τα 20 δις. Και ω προ τη μελέτη αντικτύπου που από ό,τι φαίνεται έχει εκπονηθεί, ήθελα να καταλάβω ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεδομένου του μεγάλου αντικτύπου που θα υπάρχει στη γεωργική οικονομία. Η κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Εγώ θα πάω σε ένα άλλο θέμα Πέρυσι είχαμε την στρατηγική για τα δάση είχαμε μια πολύ ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Είχαμε μιλήσει για την αποδοτικότητα των πόρων και ότι θέλουμε την ε, ε, ε, χρήση τη σταδιακή των ε, μέσων και ήταν ξεκάθαρο ε, βέβαια ότι δεν ξέραμε ποια είναι τα μεμονωμένα μέτρα. Τώρα θέλω να ρωτήσω ε, πώς βλέπετε την εφαρμογή από την πλευρά της Κομισιόν αυτής της ευρείας στρατηγικής και έχετε λάβει υπόψη τα σημεία του Κοινοβουλίου που είχαν ψηφιστεί με τόσο μεγάλη πλειοψηφία ε, με βάση την αποδοτικότητα των πόρων και ε, φυσικά σε σχέση με τα υποχρεωτικά κριτήρια για τη βιομάζα που θα έχουμε στο μέλλον. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν η γνώμη σας και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή μας ε, για ε, τις περικοπές στην Αυστρία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ουγγαρία. Ε, έχουμε ε, μαζικές φυσικές καταστροφές εκεί και θα ήθελα να το έχετε και αυτό κάπου στο μυαλό σας όταν γίνονται κάποιες προτάσεις για αυτά τα κράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμπληρώσω αυτά που είπε και η συνάδελφος. Ε, καταρχάς ε, για τη γραφειοκρατία. Ε, κύριε Επίτροπε, το αναφέρατε, αλλά κάπου χάνετε το μήνυμα. Είπατε για μια προκαταρκτική μελέτη για να φύγουν οι υπερβολικοί κανονισμοί στην ε, γεωργία έχουμε ε, μία ε, απέτηση για ένα τετραγωνικό, δηλαδή 30 cents και καταλαβαίνετε ότι όλοι σε εσά θα προσφεύγουν στην Γερμανία ε, και θα πηγαίνουν προς τις Βρυξέλλες και ούτω καθεξής. Ε, τώρα για το τεμήνιμις είπατε ότι θα υπάρξει μείωση των αποθεμάτων στα κράτη-μέλη ε, έτσι ώστε να φτάνουν τα μέσα για, των ζωοτροφών που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Κύριε Άγνιο, θέλετε πάλι το λόγο. Όχι, όχι. Ωραία. Οπότε εξαντλήσαμε το κατάλογο των ομιλητών. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και πώς μπορεί να επιβαρύνει τους γεωργούς Θα ήθελα και αυτό να το σχολιάσετε. Και έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ε, υπευλήθησαν πολλές ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Παρακαλώ, περιμένουμε τις απαντήσεις. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις και σας ευχαριστώ όλους. Για τις ερωτήσεις σας Πολλοί ρωτήσατε για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Το ανέφεραν πολλοί. Είναι σημαντικότατο ζήτημα για τι συμφωνίε ελευθερών εμπορίου όπως συνάψαμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν διαφορετικό σύστημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Και για την προστασία των γεωγραφικών περιοχών. Πρόσφατα αντιμετωπίσαμε μεγάλη δυσκολία για να αναγνωριστεί αυτή η πραγματικότητα. Ω διαπραγματευτή όμως, νομίζω ότι πραγματικά βρήκα ένα παράθυρο ευκαιρία ώστε οι ΗΠΑ να κατανοήσουν έστω τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων και του συστήματό του για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να του πείσουμε ότι μπορεί να βρεθεί συμφωνία ε, εντό τη TTIP. Εάν το πετύχουμε θα είναι καλό αυτό, εάν συμπεριλαμβάνονται γεωγραφικέ ενδείξει. Σα διαβεβαιώ λοιπόν και εσά και όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται για τι γεωγραφικέ ενδείξει, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Όλα τα κρατη έχουν κάτι να κερδίσουν από αυτό. Και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στι γεωγραφικέ ενδείξει. Εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ικανοποιήσουν τι απαιτήσει μα για τι γεωγραφικέ ενδείξει, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Τέρμα. Ω προ την αρπαγή γεών. Η κυρία Χάουσλινγκ νομίζω ότι ανέφερε το Η κυρία Χόιμπους μάλλον. Μιλήσατε για την ε, σύγκριση με βάση τα εκτάρια μεταξύ των χωρών και των ε, περιφερειών. Όμω δεν μπορούμε να έχουμε ακριβεί πληροφορίε όπω για την έκταση των ε, περιοχών, την επιφάνειά του, τη σχέση αγοραστών και πολιτών. Αυτό είναι κάτι που τα κρατη μέλη μόνο μπορούν να το καταγράψουν. Μπορούμε εδώ να μιλάμε για επικουρικότητα, πολλοί το συζητάνε εδώ, αλλά τα κάτι μέλη και οι περιφέρειέ του, οι περιοχέ του, εκείνε συλλέγουν τα ακριβή δεδομένα. Η Eurostat έχει δημοσιεύσει κάποια στοιχεία για τις ε, γεωργικές τιμές ε, το, από το 2009 για τις γεωργικές τιμές και την τιμή των διαφόρων εκτάσεων. Εάν θέλουμε να βρούμε μια κοινή μεθοδολογία για να γίνουν τέτοια στατιστικά ε, συλλογή τέτοιων με δεδομένων που να είναι συγκρίσιμα, μπορούμε. Αλλά η Eurostat μέχρι το τέλο τη χρονιά θα, θα δημοσιεύσει κάποια στοιχεία, καλύπτοντα την τελευταία πενταετία για τι σχετικέ τιμέ. Γενικώ πάντω, οι πληροφορίε που μπορώ να σα δώσω έχουν να κάνουν με τι τάσει που επικρατούν. Όχι όμω με συγκεκριμένη φωτογραφική παρουσίαση των δεδομένων. Όσο για το μέλι. Και το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ. Στο πρόγραμμα των στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων δεν το θίξαμε αυτό το πρόγραμμα ακόμα. Δεν συμπεριλαμβανόταν στην εντολή. Οι πορτογαλικές αρχές θα έπρεπε να το λάβουν υπόψη ε, για τη βελτίωση της εντολής εφόσον θέλουν να ασκήσουν ε, κάποια επιρροή και για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Εάν η παραγωγή από την άλλη θέλουν να παράγουν περισσότερο γάλα για χαμηλότερε τιμέ, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε προ στιγμή. Ε, δεν προέβλεψα εγώ την κατάσταση αυτή συμφωνήθηκε από τους νομοθέτες εδώ το 2003 και 2008 και το 2013. Έχουμε σαφώς μια τρικυμία εδώ με παγκόσμια υπερπαραγωγή, υπερβολική προσφορά. Κανεί δεν το είχε προβλέψει αυτό το 2003. Ότι στην αγορά στι ΗΠΑ λόγω χάρη στην Αυστραλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα θα υπάρχει υπερπροσφορά. Ε, μαζί με την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και έχουμε μια ευκαιρία με το άρθρο 222, με τις ε, αποσυνδεδεμένες κριτικές βοήθειες. Υπάρχει μάλλον εκεί με την ε, δυνατότητα αυτή της, του διπλασιασμού των κρατικών βοηθειών και της εξελαχής των όροφες που ισχύουν την τελευταία διετία, να καταφέρουμε μερικά πράγματα σε κριτικό επίπεδο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να βρούμε λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πρέπει να τα δούμε σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να τα δουν οι γεωργοί και οι παραγωγοί. Είναι θέμα των ίδιων των γεωργών ή των παραγωγών. Και να δούμε τι βοήθεια μπορούν να λάβουν από την ε, βοήθεια των, ε, από τις κρατικές βοήθειες. Και εσείς αναφέρατε τις γεωγραφικές ενδείξεις για τη σχετική συμφωνία. Μιλάμε για την συμφωνία με τον Καναδά εδώ. Νομίζω ότι η συμφωνία ήταν αρκετά καλή, ήταν ισορροπό το αποτέλεσμα και θα τα δούμε, θα τα συγκρίνουμε εφόσον χρειαστεί. Κυρία Χάουζεκαμπ, για το κλίμα και την βιολογική Γεωργία. Έχουμε πολύ καλή σχέση συνεργασία με τον κύριο Βέλα, τον υπεύθυνο για τα θέματα αυτά του κλίματος Και επανειλημμένω έχουμε συζητήσει το τι γίνεται για το νερό, τη βιώσιμη εντατικοποίηση της Γεωργίας και ελπίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Βήματα προόδου στο εγγύς Για τα οικοσυστήματα, την αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στο γεωργικό σύστημα, σας διαβεβαιώ όλους εδώ ότι πραγματικά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και στο σωστό κλίμα σκέψεις ε, για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε για τη Γεωργία. Ο κ. Νταντά ανέφερε τα θέματα τα θέματα ανταγωνισμού. Ξέρετε ότι εδώ έχουμε κατευθυντήριε γραμμέ τι οποίε με την Επίτροπο Βέσταγκερ είχαμε επεξεργαστεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο ανταγωνισμό και η γεωργία μπορεί να μην είναι βρίσκονται ακριβώ στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή, αλλά θέλουμε να υπάρχει συνέπεια. Συνέπεια σε όλε μα τι πολιτικέ, με συστηματική τακτική αναθεώρηση από τι αρχέ ανταγωνισμού των καταμελών. Και όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει έκθεση, έλαβε έκθεση που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο το 2012, το οποίο η οποία επεσήμανε σημαντικέ αποκλήσει στι πρακτικέ μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού των διαφορών καταμελών, την, την αναλύσαμε διεξοδικά. Για να μην πω υπερβολικά καταληπτό, ένα για το τι ισχύει στην αγορά και δεύτερον για το τι πρακτικέ έχουν ε, η παραγωγή και τι κυρώσει επιβάλλονται από τι εθνικέ αρχέ. Το αποτελέσμα ήταν τα περισσότερα μπορούσε να τα εξηγεί κανεί με τι διαφορετικέ ε, εθνικέ καταστάσει. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί να ανοίγει άλλη σειρά απορριών. Ε, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πω την άριστη συνεργασία μα. Συνεργασία μεταξύ Επιτρόπου Ανταγωνισμού και Επιτρόπου υπεύθυνο για το άρθρο 222. Πρόσφατα επικαλέστηκε και εκείνη το άρθρο 222. Αυτό είναι καλό. Οπότε ασχέτω των εξαιρέσεων από κάποια μέτρα ανταγωνισμού, ο ανταγωνισμό. Επίτροπε. Ε, ο ανταγωνισμός ε, ω τώρα στην Επιτροπή ήταν πολύ χρήσιμο και για τα δικά μα θέματα. Κύριε, κύριε Τάκουλα για τη Φινλανδία. Έτσι γίνεται με τι υποκαταβολέ και το επίπεδο του 70%. Πάντω λαμβάνω υπόψη αυτά που είπατε, ότι μερικά κράτη-μέλη μπορεί να αποφάσισαν, να το κάνουν αυτό αν είχαν περισσότερο χρόνο. Ίσως μέχρι το τέλο τη χρονιά να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Πρέπει να, δείξουμε, να ρίξουμε μια ματιά στην Φινλανδία. Έχω δώσει παράταση για του ετούντε. Για τα σχετικά προγράμματα. Θα πρέπει όμω οι περιφέρειε των κρατών μελών να δουν αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα. Κάποιοι πρόσωποι των περιοχών, ομών, επαρχιών είπαν ότι δεν είναι αρκετό χρόνο μέχρι 15 Μαου. Του δώσαμε λοιπόν ένα μήνα μέχρι 15 Ιουνίου. Η Ρουμανία τώρα. Κι άλλοι. Γαλλία. Και μερικέ περιοχέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει θέμα με αποπληρωμή των ποσών που εκκρεμούν από το 2015 λόγω προβλημάτων στο σύστημα πληροφορική. Θα τα δούμε αυτά Τι ερχόμενε ημέρε. για να δούμε αν μπορούμε να διευκολύνουμε τη Ρουμανία χωρίς να επιβληθούν τιμέ και πρόστιμα. Ποινές και πρόστιμα. Διότι ο στόχο δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να τιμώρει τα κράτη-μέλη. Επικρατεί η κοινή λογική εδώ Και δεν θέλουμε να κατηγορείται η δημοσιονομική διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με αυθαίρετους ελέγχου ε, και περιοχέ ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καταφέρουν να δαπανίσουν τα ποσά που του αναλογούν. Είμαι βέβαιο ότι οι αρχέ θα τα αντιμετωπίσουν σωστά και θα επιληφθεί το πρόβλημα. Επίση, ρωτήσατε τι γίνεται με όλου αυτούς τους ανθρώπους που δεν δαπανούν τα ποσά που του αποδόθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Νομίζω πολύ. πολλά μάλλον μέλη Οκτώ συγκεκριμένα γνωρίζουν τέτοιε περιπτώσει. Καταλαβαίνω ότι έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια είναι. Τα κράτη-μέλη που δεν έχουν δαπανίσει τα ποσά είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Κύπρος, οι κατοχώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Φιλανδία. Έχουν μέχρι το τέλος Ιουνίου για να τα δαπανίσουν. Η απάντηση είναι ανασκουμποθείτε. Και άλλες χώρες έχουν κρέμια ποσά. Πραγματικά με ευνηδιάζει αυτό σε αυτή τη φάση που δεν έχουν ακόμα ξοδέψει τα χρήματα όλοι αυτοί. Είναι δύσκολο να τους δίνεις χρήματα και να μην τα ξοδεύουν. Ως προς την ζημία από τους παγετούς. Είτε πρόκειται για τα αμπέλια είτε για άλλες καλλιέργειες. Την περασμένη μόλις εβδομάδα εκδόθηκε μια σχετική σύσταση για την Κροατία. Θέλουμε να υπάρξει κάποια διαλεκτικότητα, ίσω με το πρόγραμμα τη ανάπτυξη τη υπαίθρου να προβλεφθούν πρόσθετα μέτρα για να στηρίξουμε την Αυστρία, την Κροατία, την Νότια Γαλλία και άλλε χώρε, τη Σλοβενία, ξέρω εγώ, για τα θέματα αυτά. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σε μια ερώτηση για την οποία μόλι έλαβα την ε, τεκμηρίωση τι προηγούμενε ημέρε. Το γνωρίζουμε όμως και τα είπε και ο υπουργό σας στο περασμένο Συμβούλιο. Κύριε Κούσμιο, σας ε, συγχαίρω για την εκλογή σας στη θέση του Αντιπρόεδρου. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα για την Πολωνία. Και θέλουμε να μην υπάρχουν δεσμολογικοί φραγμοί για τα και μήλα και ιδίω την αποστολή του στι ΗΠΑ, υπάρχει εκεί μια διαδικασία διαβούλευση που δεν θα επιτρέψει να καλυφθεί η σοδειά σα το 2016, αλλά ελπίζουμε ότι το 2017 μπορεί να έχει επιληθεί το θέμα. Έχουμε πάντω πετύχει να σα βρούμε νέα ανοίγματα στην αγορά τη Ιαπωνία. Σα αφορά και αυτό, Πολωνία. Είναι λοιπόν καλή κατεύθυνση που έχει πάρει η, η όλη υπόθεση. Είσαστε μεγαλύτερη παραγωγή μήλων στην Ευρώπη, η Πολωνία. Πολλοί από εσά είπαν ότι αν δεν έχουμε χρήματα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να καταφύγουμε στο Ταμείο Αντιμετώπιση τη Κρίση. Δύσκολη ερώτηση, αλλά ήθελα να ακούσω τι απόψει κάποια στιγμή. Διότι εάν επισυμβεί κάποια κρίση σε έναν από του βασικού μα τομεί παραγωγή, θέλουμε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια συνετή οικονομική απάντηση. Για την τροφική αλυσίδα, την αναφέρατε πολύ. Νομίζω η κυρία Μαρτίνε επίση την ανέφερε για την Ισπανία. Έχουμε προβλήματα στη Γαλλικία. Υπάρχουν εθελοντικές ε, συνδεδεμένες βοήθειες αναγελάδα για τους γαλακτοπραγωγούς ε, στην Ισπανία. 200 ευρώ αναγελάδα. Πολλοί θα θέλαν τα να έχουν τέτοιου είδους λύσεις. Έχουμε θέματα ζωικής ευζοίας. Αλλά υπάρχουν και δικές σας εθνικές αρχές που μπορούν να καλύψουν τα ζητήματα της ε, ευζοίας των ζώων. Εμείς έχουμε ε, ευθύνη ως νομοθέτες ε, και επίσης έχουμε μεγάλες ευθύνες για τη διαχείριση του προπολογισμού. Ως προς τη διαλεκτικότητα και την ευελιξία που προσφέρουμε σε τομεί σε συγκεκριμένε περιοχέ για να ανταποκριθούν στην κρίση, προφανώ και προβλέπεται. Αλλά πρέπει να τα πάμε καλύτερα, όπω λέτε και εσεί, στο πρόγραμμα ανάπτυξη τη υπαίθρου, για να μπορούμε να μετακυλήσουμε τα κονδύλια από το ένα πλέον στον άλλο, εφόσον χρειάζεται σε περίπτωση κρίση. Στου τελευταίου έξι μήνε πρέπει και εσεί να κοιτάξετε πώ θα μεταρρυθμίσετε το πρόγραμμα σα για την ανάπτυξη τη υπαίθρου, ώστε να αντιμετωπίσετε καλύτερα αυτέ τι έκτακτε ανάγκε. Πάντω, στα κράτη-μέλη πρέπει να υπάρχουν εύκολη αναθεώρηση τέτοιων προγραμμάτων για να αντιμετώπιση των περιπτώσεων κρίσεων. Ξέρω τι κάνουν οι δικέ μου αρχέ και σε ποιο χρονικό πλαίσιο σε ανάλογε περιπτώσει. σω τα κάτι μέλη να μην τα γνωρίζουν όλοι. Ω προ τον κύριο Ντεβάιλο και την Πορτογαλία, βεβαίω ε, το θέμα των παραγωγών είναι κάτι που μπορούν να διαθετήσουν ε, ε, τα κάτι μέλη, όμω δεν έχει κανένα λόγο να απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αναδιάρθρωση. Ε, το προβλέπουν οι κανόνε, τα στοχευμένα μέτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τι κατοικέ βοήθειε, τι οροφέ εξυλαχή αλλά δεν μπορούμε να μαντέψουμε περαιτέρω τι θα κάνουν τα δημοσιονομικά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τους μεμονωμένους παραγωγούς και το τι οικονομικέ επιπτώσει θα έχει για την κοινότητα των γεωργών σα η προσπάθεια αναδιάρθρωση, για τη γεωργία και το εμπόριο. Κύριε Καπούτο, σωστά τα είπατε. Οι συνέπειε των συμφωνών ελεύθερων συναλλαγών είναι κάτι που πραγματικά με αποσχολεί. Θα έχει περατωθεί σχετική μελέτη μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα έχουμε μια πιο ε, μια πιο απτή θέση για το τι περιθώρια έχουμε για τι κινήσει μα για το μέλλον. Αναφέρετε τη Μερκοσούρ. Είναι πολύ σημαντικό που ο Υπουργό σα Γεωργία και ο Υπουργό Εμπορίου σα συζητούν μεταξύ του. Μπορεί να μην συμφωνούν πάντοτε στα θέματα αυτά, να μην ταυτίζονται οι απόψει του, αλλά συζητούν τουλάχιστον. Αυτό ισχύει και για άλλα κρατημέλη. Πάντω υπάρχει συντονισμό μεταξύ Υπουργείων. Κάτι είναι και αυτό σε δύσκολου καιρού. Και εξαρτάται και από το επιμέρου ζήτημα κάθε φορά. Όμως νομίζω ότι η Μερκοσούρ είναι ένα κλασικό παράδειγμα όπου θα πρέπει το εμπόριο και η Γεωργία να συζητούν σταθερά. Για κάθε δασοκομεία και τα δάση. Προωθούμε τα βιώσιμα δασικά προϊόντα, την βιολογική οικονομία, την βιοενέργεια ναι, η στρατηγική μα για τη είναι κάτι που μα απασχολεί τακτικά με εφαρμοστικά προγράμματα για να λάβουμε απόψη ακριβώ το τι προβλέπει η συνολική μα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δοσοκομεία. Ευχαρι... Συμφωνούμε κύριε Ροπέ. Έχουμε γαλακτοπαραγωγού όλα τα κάτι και μπόρεσα να κάνω κάτι συγκεκριμένο για τα βαλτικά κράτη, τα κράτη τη Βαλτική στην αρχή τη θητεία μου. Αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει και σε άλλα κατημέρια, Όλοι έχουν πρόβλημα με του γαλακτοπαραγωγού του. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιο τρόπο μεταξύ των εργαλείων που έχουμε στο κουτί μα να δούμε τι θα γίνει με μια ευρωπαϊκή απόκριση. Αλλά η α, συγκεκριμένη λύση δόθηκε στοχευμένα για τα κράτη τη Βαλτική. Δεν μπορεί να δοθεί και για του υπόλοιπου η ίδια. Συμφωνώ πάντω μαζί σα. Θα ήταν καλό εσεί ο ίδιο να συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό σα, τον Υπουργό σα και του ενδιαφερομένου και να σκεφτούμε το κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρχουν 23 διαφορετικά σύνολα μέτρων. Ελπίζω η αγορά να σταθεροποιηθεί και να βελτιωθεί στο μέλλον. Και έχω αναγνωρίσει την έλλειψη ε, των, ε, ε, κύριε Φλάναγκαν, ίσως να μην ήσασταν εδώ. Αναγνω, το αναγνώρισα. Στις αρχές του 2015 δεν θα ήσασταν εδώ, γιατί την αναγνώρισα Δεν είπα τίποτα για αυτό το θέμα. Είμαι... Χαίρομαι που είναι καλά. Πάντω 50.000 τόνοι παραπάνω από την παραγωγή γαλακτό. Ε, κοιτάξτε, εγώ το είπα, το ανέφερα, επιλέξει, διότι υπήρχε κρίση. Το έχω πει στι αρχέ του 2015. Τώρα ήσασταν εσεί εδώ ή όχι, δεν το ξέρω. Ήμουν, ε, το είπα. 5.000 τόνοι παραπάνω. 50.000 τόνοι παραπάνω. 150 εκατομμύρια τόνοι παραπάνω γάλα στην Ευρώπη. Γι' αυτό υπάρχει πίσω στι τιμέ και γι' αυτό πρέπει να βρούμε ένα μαξιλαράκι στην αγορά. Ε, γι' αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στήριξη. Απλούστευσα τα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου προκειμένου να επιτρέψουν στα κατημέλη να μπορέσουν να τροποποιήσουν τα προγράμματά του. Τουλάχιστον τα ετησίω και να μπορούν να μετακυλίουν τα κονδύλια εφόσον το θέλουν. Αλλά δεν είμαι υπουργό τη Ιρλανδία ούτε πουθενά αλλού. Θα πρέπει οι ίδιοι να τα αλλάξουν αυτά και να υποβάλουν τα αιτήματά ε, του. Και εντό ευλόγου χρονικού διαστήματο. Συμφωνώ ότι χρειάζεται ευελιξία και διαλλακτικότητα. Τώρα τι θέλετε να σα πω, τι θα γίνει με τον Brexit. Εγώ και ο κύριο Άγνιο είχαμε μια υπέροχη συζήτηση πρόσφατα και καλό ήταν να, σας να σα παραπέμψω σε αυτήν. Ήταν πολύ διασκεδαστική κιόλα. Κυρία Μίλλερ, για την Ουκρανία και την όλη συζήτηση. Είναι σημαντικό να έχουμε εμπορικέ ε, διαπραγματεύσει γι' αυτό, αλλά μόνο οι γεωργοί έχουν ε, υποστεί τι συνέπειε των ε, αποφάσεων τη κοινή αγροτική πολιτική. Δεν μπορώ να μαντέψω τι θα γίνει μακρά, πιο μακριά στο μέλλον για τα θέματα αυτά. Ο υπουργό σα θα τα ξέρει καλύτερα. Το ίδιο και ω προ την αλληλεγγύη που εκφράστηκε για την εισβολή σε ένα τμήμα τη Ουκρανία. Καταλαβαίνω τι έχει γίνει αλλά εν τέλει οι ρωσικέ αρχέ αποφασίζουν να επιβάλλουν εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα. Δική του απόφαση είναι. Ε, Εμεί προσπαθήσαμε ακόμη και μέσω του Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξομαλύνουμε τι σχέσει, ε, ιδίω τα γεωργικά με τον κύριο Πούτιν, αλλά εκείνο δεν δεσμεύτηκε για τίποτε. Χρειάζονται δύο για να χορέψει κανεί ταγκό και δύο για να βρεθεί συμφωνία. Ε, προσε... σημειώνω ότι κάποιοι μιλούν πολύ για τα χρήματα της ΚΑΠ, για τα ποσά που διατίθεται στην ΚΑΠ. Ο Γερμανός Υπουργός τουλάχιστον μίλησε για 10% περικοπές στα ευρωπαϊκά προγράμματα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων. Πρέπει να τα δείτε και λίγο έτσι. Προσπαθούμε να εξορροπήσουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά στην ε, ε, ατζέντα μας. Δίνονται προτεραιότητες σε κάποιες πολιτικές καταφορές εναντί άλλων η δυνατότητα λιγμών είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ό,τι κάναμε προηγουμένως για την παραγωγή και το τι κάνουν οι νεαροί γεωργοί. Πρέπει να σπρώξουμε περισσότερους νέους και να τους παροτρύνουμε να ασχοληθούν με τη γεωργία. Ε, αλλά θέλουν να αισθανθούν οικονομική ασφάλεια για να κάνουν κάτι τέτοιο και να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίε. Χρειάζονται πάλι λοιπόν και άλλες πολιτικές για να το πετύχουμε. Για τις κλιματικές αλλαγέ, Πρόεδρε είτε σας αρέσει είτε όχι, οι κλιματικές αλλαγές θα είναι αναπόσπαστο τμήμα των πολιτικών πρωτοβουλειών μας στο μέλλον. Η Διεθνή Συμφωνία στο Παρίσι, τις οποίες τμήμα θα και η Γεωργία, ως προς τις πολιτικές που προτείνονται από, την, από τον Επιτροπο Καρνιέτε, και επειδή ήταν στο Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και εκεί τόνισε ότι η Γεωργία θα πρέπει να παίξει το δικό της ρόλο για τη μείωση των εκπομπών, Αυτά λαμβάνονται υπόψη. Οι πολιτικέ μα στο μέλλον θα, θα επηρεαστούν από τι διεθνεί συμφωνίε. Η βιωσιμότητα στη Γεωργία είναι κάτι που θα παραμείνει σταθερό. Η βιωσιμότητα στη Γεωργία για τι πολιτικέ για τι κλιματικέ αλλαγέ και το περιβάλλον θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο οποιοδήποτε πολιτική πρωτοβουλία θα υποβληθεί από την Επιτροπή στο μέλλον. Κυρία Πέρικ, αναφέρετε και εσεί τη Ρωσία, αλλά και το αποθεματικό για την κρίση. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα σκεφτείτε μόνοι σα. Εσείς θέλετε να υπάρξει στήριξη. Θέλετε ένα τέτοιο χρηματικό πακέτο για το μέλλον. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ μόνος μου. Κυρία Γκαρσία, να πω ότι οι φήμες για το πρόγραμμα ανάπτυξη της υπαίθρου ήταν ε, ατελείωτες στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή οι φήμες φαίνεται να μην μπορούν να ρίξουν σκιά στο πρόσωπο του νέου προγράμματος για, για το, για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι πολλέ οι περιοχέ που ωφελούνται από αυτό και υπάρχει και μεγάλη ευελιξία στα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου καθώ και προσπάθεια απλούστευση. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Έχουμε μια συνάντηση τη ομάδα υψηλού επίπεδου με τον Επίτροπο για την Ανάπτυξη τη Υπαίθρου και την Απλούστευση, την κυρία Κρετσού, ε, η οποία θα ασχοληθεί ακριβώ με αυτό το θέμα. Το ζήτημα των ε, αρχών της αγοράς και της ίδρυσης παρατηρητηρίου για το γάλα χείρι προχωρήσει, θα γίνει κατά ανάλογα το πρόγραμμα και το χείριο. Είναι σημαντικό αυτό μήνυμα και προ την αγορά. Ακούω λέτε για τα προκυπευτικά, αλλά δεν θα προβλέψουμε μια νέα τοποθέτηση. Η παρέμβαση στις τιμέ αναφοράς και τις τιμέ τη αγορά για τα προκυπευτικά ε, είναι κάτι διαφορετικό δεν ε, μπορούμε παρά να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του ρωσικού εμπάργου. 75% των προκυπευτικών μας βρέθηκαν, βρήκαν νέα ανοίγματα στην αγορά. Βρήκαμε λοιπόν τρόπο να στηρίξουμε την αγορά προκυπευτικών και να προστατεύσουμε το όλο σύστημα από το ρωσικό εμπάργο. Η τέλεια λύση δεν έχει βρεθεί, αλλά δεν υπάρχει ακόμα και πλήρη συμφωνία για το μέλι. Δεν είμαι και πολύ πυρογνώμων για το μέλι, ομολογώ. Ο κύριος Σέρντος μίλησε για την ε, μεγαλύτερη δηματοληψία στα εξωτερικά σύνορα για το μέλι. Αλλά αυτό είναι θέμα και αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Σάντετε για την υγεία. Θα διαβιβάσω πάντως τα σχόλιά σας στον συνάδελφο Επίτροπο Αντρίου Κυρία Ντότς, είπατε ότι δεν ε, μπόρεσα να πάω στη γεωρική έκθεση, αλλά ε, ξέρετε ότι συνάντησα πολλούς Γιώργους, γιατί πήγα σε αγρόκτημα και είμαι εξοικειωμένος με τα θέματα που ε, επισημάνατε. Και πριν την έκθεση ε, μίλησα εκτενώς με τους Γιώργους της ε, περιφερειάς σας. Ήταν πολύ επικοδομητικές συζητήσεις και ακολούθησε και αλληλογραφία. Σε ό,τι αφορά την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, κυρία Τότς. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για το κατά πόσο θέλουμε ε, κάτι τέτοιο και τι θα συμπεριλάβουμε σε αυτή. Έχουμε ε, επιλογή είτε για μικρές αλλαγές είτε για πιο ουσιώδη και ε, πιο βαθιά ενδιάμεση αναθεώρηση. Αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει τι είδου αναθεώρηση επιθυμούμε. Και τι επόμενε εβδομάδε θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά για το τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε των μικροαλλαγών ή των πιο ρηξικέλευθων τροποποίησεων. Ε, ελπίζω να μην άφησα κανέναν παραπονεμένο. Προσπάθησα να καλύψω όλες τις ερωτήσεις και σας ευχαριστώ για την πληθώρα των ερωτήσεων που υποβάλλατε. Ε, και φαντάζομαι ότι και στο επόμενο πρόγραμμα εργασία για το 2017 θα συμπεριλάβουμε πολλά από αυτά που είπατε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Φλάναγκαν, παρακαλώ, εν συντομία. Ε, σχολιάσετε την παρουσία μου στις συνεδριάσεις. Μπορεί να μην σας αρέσουν αυτά που λένε όταν έρχομαι, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος που έρχεται τακτικά στην Επιτροπή θα μπορούσε να πει ότι δεν είμαι πάντα εδώ. Και τα σχόλια σας για την προσέλευση μου ε, συνέπειτα με την εποχή που απουσίαζε, επειδή ήταν πολύ βαριά στη η γυναίκα μου. Το γνωρίζετε, αλλά παρόλα αυτά δεν χρησιμοποίησατε αυτή την προσωπική ε, προσβολή. Αυτό πραγματικά είναι ντροπή, ξεδιάντροπο. Ε, Ούτω ή άλλω είχα κακή γνώμη για εσά, αλλά μετά από αυτό πραγματικά πέσατε πάρα πολύ χαμηλά στα μάτια μου. Είναι αειδιαστικό, είναι ξεδιάντροπο αυτό που κάνετε. Με συγχωρείτε να απαντήσω. Δεν είχα καμία γνώση της ασθένειας της σύζυγου σας. Δεν το γνώριζα. Δεν διαβάζω εφημερίδε καθημερινά. Με συγχωρείτε, ούτε τα θυμάμαι και κιόλα μετά. Δεν διαβάζω καν αυτέ τι εφημερίδε. Αλλά αν είστε τόσο ευαίσθητο για αυτό το θέμα, που δεν είσαστε εδώ όταν μίλησα για ένα θέμα πολιτική, που δεν είχε καμία σχέση με την προσωπική σα ζωή, καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι δεν είχα μια πρόθεση να σχολιάσω τα προσωπικά σα. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ, μην μεταφέρετε τα εθνικά σας προβλήματα εδώ στην Επιτροπή μας. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι ήταν μια πολύ σοβαρός ε, και φιλικός διάλογος μεταξύ πραγματικών εταίρων. Πολύ καλή οργάνωση και προετοιμασία και αυτό περιμέναμε από ένα διαρθρωμένο διάλογο. Ε, ίσως μερικοί θα θέλαμε να ακούσαμε περισσότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που έγινε αυτός ο διάλογος μεταξύ πραγματικών εταίρων. Είναι οι ιδιαίτερες οι περιστάσεις αυτή τη στιγμή στη Γεωργία. Έχουμε το ρωσικό εμπάργο, έχουμε το TTIP, ε, τις επικείμενες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Ειδικέ περιστάσεις ε, που επηρεάζουν και τη γεωργία. Αυτή είναι η κατάσταση. Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν και τη γεωργία. Και φοβόμαστε για το μέλλον της γεωργίας ε, στη συνέχιση των ε, διεθνών διαπραγματεύσεων για διάφορες συμφωνίες. Ε, είτε το θέλουμε είτε όχι, κάποιο εξορθολογισμός πρέπει να γίνει στη γεωργία. Και αν τα κρατημέλη είναι υπέρ τη κοινή γεωργική πολιτική ε, είναι γιατί το κάνουν ε, έχοντας επίγνωση και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά ε, τηρώντας τους, ε, τις αρχές του δίκαιου ανταγωνισμού, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των συνθηκών και ο θεματοφύλακας και του θεμητού ανταγωνισμού και φροντίζει για τις ε, όρους θεμητού ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά το, την κατάσταση στην ε, Ισπανία. Το πρόβλημα της κατακόρυφης ολοκλήρωσης, ε, της αποτελεσματικότητάς της και της σωστής οργάνωσης ε, δεν είναι αδιάφορο με τις τιμές. Έχει κάποια σχέση και με τις τιμές τις γεωργικές. Και σίγουρα ένα αποτελεσματικό σύστημα επηρεάζει και πλήττει και τους Σε ό,τι αφορά τώρα αυτές τις εκούσιες συμφωνίες για το θέμα της, του περιορισμού της παραγωγής. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η εκούσια ε, συμφωνία για τον περιορισμό της παραγωγής. Θα πρέπει να έχουμε κάποια ε, κάποιους μηχανισμούς παροχής κινήτρων, εναυσμάτων και ίσως ε, και κάποιες ενισχύσεις για τον περιορισμό της παραγωγής. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για το γάλα, για παράδειγμα, γιατί έχουν δάνεια οι κτηνοτρόφοι, η γαλακτοπαραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε και οικονομικά κίνητρα, αν θέλουμε μείωση της παραγωγής και πιο αποτελεσματική διαχείριση. Και εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με τις μεγάλες αλυσίδες διανομής τροφίμων και την τροφική αλυσίδα. Ήταν αρκετά εκτενή συζήτηση, κράτησε πάνω από δύο ώρες. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Επίτροπη και ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήρθαν συνοδεύοντας τον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ. Ε, ένα λεπτάκι διακοπή για να ξεπροβοδίσουμε τον Επίτροπο και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Αρμόδια ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ενώ εμείς θα εκπονήσουμε γνωμοδότηση το θέμα. Το έχει αναλάβει η κυρία Βιόριτσα Ντάντσιλα. Πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Και κρίναμε σκόπιμο να αναλάβουμε αυτή τη γνωμοδότηση για να εξοικειωθούμε με το θέμα. Θα ήθελα πρώτα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα κάνει την παρουσίαση και κατόπιν θα δώσω το λόγο στη συντάκτρια γνωμοδότηση, την κυρία Νταντσίλα. Ο κύριος ε, Φιλίπ Μαγκνέ ε, από Στην τελευταία συνεδρίαση μιλήσαμε μαζί του από το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας. Ε, είχε πει ότι θα έρθει. Α, δεν έχει έρθει ακόμη. Οπότε, ας δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο 6. Περιμένουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει το λόγο, την εκπρόσωπο μάλλον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας ε, αποστήλατε για να κάνουμε μια παρουσίαση. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, και ε, έχω συγκεκριμένη επικέντρωση στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην αγροτική ανάπτυξη. Αν δείτε την παρουσίαση θα δείτε μια γενική επισκόπηση της έκθεσης του άρθρου 16 που είναι μια συγκεκριμένη υποχρέωση που έχουμε στον κανονισμό να δείχνουμε τα αποτελέσματα ε, για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και την νεολαία και θα δώσω συγκεκριμένη προσοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Νομίζω ότι ε, πρέπει να ξεκινήσω με τα χρήματα. Ε, για το 2014 μέχρι το 2020 έχουμε 454 δις ευρώ στα ταμεία αυτά. Αν βάλουμε και την εθνική συγχρηματοδότηση, ε, φτάνουμε στα 627 δις. Το κομμάτι του ε, τα είναι 29 ε, δις από το πρώτο ε, ταμείο, δηλαδή 4 δις από το πρώτο πυλώνα και αν δούμε και τα top-up έχουμε 161 δις για αυτό το ταμείο που είναι σημαντικός προϋπολογισμός. Αν πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε λίγο τα νούμερα για να καταλάβετε την σημασία των διαφορετικών και επενδυτικών ταμείων σε επίπεδο επενδύσεων. Βλέπουμε τη συνολική δημόσια επένδυση, είναι και αυτό κομμάτι της έκθεσης άρθρου 16 και βλέπουμε εδώ ότι ε, έχουμε 14% της, ε, των ε, δημόσιων επενδύσεων που προέρχονται από αυτά τα ταμεία, όμως για την Πορτογαλία, την Κροατία, την Λιτ Λετωνία, Λιθουανία και Ουγγαρία είμαστε γύρω στο 60% ε, και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι είχαμε μια μεγάλη μείωση σε σχέση με το παρελθόν, ε, το 2014, σχεδόν 80% σε πραγματικούς όρους. Αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αν δείτε την ανακοίνωση θα δείτε ότι το θέμα δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και το πώς δημιουργούμε τις σωστές συνθήκες για τις επενδύσεις. Πώς έχουμε σωστές ε, συνθήκες για αποτελεσματικό προγραμματισμό. Εδώ βλέπετε μία λίστα που ουσιαστικά δείχνει τι έχουμε κάνει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε τις εξάντε ε, αιρεσιμότητες ε, που ε, είναι πολύ συγκεκριμένες για την αγροτική ανάπτυξη και συγκεκριμένα έχουμε εκπληρώσει το 75% αλλά για τη γεωργία γενικά είμαστε λίγο πιο ψηλά σε επίπεδο εκπλήρωσης. Έχουμε μεγαλύτερο η προσοχή στα αποτελέσματα, στα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης στους προγραμματισμένους στόχους που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό. Επίσης, στα χρηματοδοτικά εργαλεία ε, την αύξηση της μόχλευσης και έχουμε ε, εισαγάγει και πολλά στοιχεία απλούστευσης όπως ας πούμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, απλουστευμένες επιλογές κόστους στα προγράμματά μας. Τώρα, το πώς θα τα αναπτύξουμε αυτά Υπάρχει μια συγκεκριμένη έκθεση που περιμένουμε αυτό το έτος. Αν πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια, εδώ ε, βλέπετε, ε, παίρνετε μια γεύση των ε, αναμενόμενων επιτευγμάτων στα αριστερά. Θα δείτε τα γενικά, έχω στα δεξιά δώσει συγκεκριμένους ε, συγκεκριμένες ε, προσδοκίες για τις ε, για τα επιτέγματα στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο μηχανογράφησης, ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έρευνας και επενδύσεων. Έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια ε, ε, εταιρείε που θα επικεντρωθούν 18,8 εκατομμύρια άνθρωποι ε, σε αγροτικές περιοχές θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μηχανογράφησης και θέλουμε να υποστηρίξουμε το 2,8% των γεωργών για να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν. Αυτό βέβαια το νούμερο περιλαμβάνει όλους τους παραδοσιακούς ε, γεωργούς, 7% ε, αυτών θα πάρουν τα χρήματα. 175.000 νέοι επίσης αγρότες ε, θα υποστηριχτούν όπως και άλλοι για να συμμετάσχουν σε σχέδια ποιότητας. Επίσης, 103 δις έχουν δοθεί για την αλλαγή του κλίματος είναι ε, η μεγαλύτερη κατανομή πόρων που είχαμε από τον προπολογισμό για αυτό το θέμα. Συγκεκριμένα για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε ε, ένα ε, συμβόλαιο 17% της γεωργικής γης και 3,5% των δασών που θα προστατευτούν στη βιοποικιλότητα. Έχουμε Επίσης ένα 15% γεωργικής γης ε, που θα προστατευτεί για το έδαφος και 14% για το νερό. 7,6% της γης επίσης ε, ε, έχει να κάνει με συμβάσεις διαχείρισης για την αποθήκευση άνθρακα. Επίσης έχουμε μια επένδυση 2,7 δις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 635.000 γεωργούς που συμμετέχουν σε ε, προγράμματα διαχείρισης κινδύνου που υποστηρίζει το Ταμείο. Το τελευταίο ε, κομμάτι της έκθεσης του άρθρου 16 έχει να κάνει με την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση. Θέλουμε να υποστηρίξουμε περίπου 2.500 εντόπιους ε, γεωργούς με το ε, leader, ε, περίπου το μισό του πληθυσμού στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε 44.000 νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν με το leader και θα έχουμε μη γεωργικές περιφερειακές επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν και αυτές 77.500 νέες θέσεις εργασίας μέσα της διαφοροποίησης με το ε, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη θέλουμε να φτιάξουμε και θέσει εργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Αλλά αυτά τα νούμερα δεν προσμετρώνται εδώ. Τελευταία διαφάνεια. Στο άρθρο 16 και στην έκθεση αυτή ε, περιλαμβάνεται και το θέμα μιας νέας ε, πλατφόρμας, ανοιχτών, ανοιχτής πλατφόρμας δεδομένων που δείχνει πώς προοδεύουμε σε επίπεδο επιτευγμάτων. Πέραν αυτής βέβαια θα έχουμε και τα κράτη-μέλη που θα κάνουν αναφορά σχετικά με την πρόοδο ε, μέσα από εκθέσεις εφαρμογής ε, που θα μας ε, οδηγήσουν σε μια κοινή έκθεση μέχρι το τέλη του έτους για τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά και Επενδυτικά Ταμεία. Πάμε πέρα λοιπόν από τα ποσοτικά δεδομένα και φτάνουμε στα ποιοτικά που θα είναι διαθέσιμα το 2017 και μέσα στα πλαίσια της έκθεσης απόδοσης των ταμείων το 2018 θα έχουμε μια άλλη ε, τέτοια αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα η συγκεκριά μας, κυρία Νταντζίλα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση που μας έκανε και ταυτόχρονα να συγχαρώ τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για την έκθεση πρωτοβουλίες που αποφάσισαν να εκπονήσουν. Θεωρώ ότι ως Ευρωβουλευτές έχουμε καθήκον Και αλλάζει μικρόφωνο η γιατί δεν ακούγονταν καλά. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση, αλλά και του συναδέλφου τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν να συντάξουν έκθεση με το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι ω Ευρωβουλευτέ έχουμε καθήκον να παρακολουθούμε την εφαρμογή. Με ακούτε. Λοιπόν, έχουμε καθήκον να παρακολουθούμε την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα η σχετική πρωτοβουλία είναι επίκαιρη γιατί ετοιμάζουμε τη ενδιάμεση αναθεώρηση του νομοθετικού πακέτου καθώς και του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Βέβαια η ανάλυση αυτή είχε προβλεφθεί για μετά από μία τριετία. Μια και όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει μόνο έτη διάρκεια, οφείλουμε να την πραγματοποιήσουμε νωρίτερα. Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων, CPR, απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο 16 να συντάξει έκθεση με την πορεία των διαπραγματεύσεων που έχει με τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πέρυσι την έκθεσή της με πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Επικεντρώμαστε σε προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και μάλιστα ο ισχύων κανονισμός απλουστεύει τα πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο και περιλαμβάνει και κάποιους στρατηγικούς στόχους, ε, αφήνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ελαστικότητα στις περιφέρειες να επιλέξουν ε, τις ε, προτεραιότητες στις οποίες θα εστιάσουν την προσοχή τους. Θα πρέπει τώρα να αξιολογήσουμε κατά πόσο η νέα μέθοδος θα ευνοήσει τη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Επίσης, καλό είναι να αναλύσουμε σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα προγράμματα εθνικής χρηματοδότησης και να, να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΑΠ. Η συνολική ε, κατανομή των πόρων από το τελευταίο Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ε, ήταν λιγότερες από, τα προηγού, από τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Αλλά σε ό,τι αφορά τα εθνικά μέτρα και την ελαστικότητά τους έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των περιφερειών. Ανάλογα με την ικανότητα του κάθε κράτους να χρηματοδοτήσει διάφορα σχέδια και ανάλογα με τις στρατηγικές επιλογές ε, των χωρών να μεταφέρουν τα μέτρα από τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ. Τα κονδύλια, ειδικά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ε, θα είναι σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του 2020 και θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για τις προσπάθειες που καταβάλουν στις διαπραγματεύσεις καθώς και την υπογραφή όλων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης ε, και μάλιστα εμπρόθεσμα. Τώρα εναπόκειται σε εμά να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση και μάλιστα την έγκαιρη χρηματοδότηση των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων και προς το σκόπο αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφύγουν να προσθέτουν απαιτήσει που ενισχύουν την περιπλοκότητα. Τέτοιες συμπληρωματικές απαιτήσει θα ενισχύσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια και θα περιπλέξει την κατάσταση. Η γνωμοδότηση εξορισμού είναι περιορισμένης ε, έκτασης και θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμπεριλάβω τα σχόλια των συναδέλφων. Θα συζητήσουμε και το θέμα αυτό μέσω μετά τις θερινές διακοπές. Οπότε και λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Ο κύριος Ροπέ, παρακαλώ, είναι ο πρώτος που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και τώρα, αλλά και στο μέλλον. Υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών, αλλά διαφορέ υπάρχουν ακόμη και εντό του ίδιου κράτου μέλου μεταξύ των περιφερειών. Βέβαια, η Ευρώπη είναι, είναι σχετικά μικρή σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον έχουμε προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Έχουμε μεγάλη αποδημία από τις φτωχότερε προς τις πιο εύπορες χώρες. Οπότε, καλό είναι να όχι μόνο να επενδύουμε σε θέσεις ε, εργασίας, αλλά να δημιουργούμε και ποιοτικέ θέσεις εργασίας, πολύ καλά αμοιβόμενες, καλύτερα από ό,τι σήμερα. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε τα φορολογικά συστήματα να ευνοούν τις περιφέρειες και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να έχουν αρκετά κίνητρα και ανάψματα για να πραγματοποιούν επενδύσεις. Στην περίπτωση της Λιθουανίας, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ατυχάνουν ε, κεντρικής διαχείρισης ε, στο Υπουργείο Οικονομίας που είναι αρμόδιο για τα θέματα αυτά. Του τέστην οι μεγάλες πόλεις λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης ενώ η ύπεθρος παραμελείται. Κάτι που δημιουργεί αστιφιλία και εσωτερικές μετακινήσεις από την ύπεθρο προς τα μεγαλύτερα κέντρα. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να έχουν περισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες και ισχυρότερη εντολή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουαζό. Στόχο ε, των διορθωτικών ταμείων και των επενδυτικών ταμείων είναι να αυξήσουν τις θέσεις απασχόληση, ε, τις επενδύσει και την ανάπτυξη στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρε. Δυστυχώ είναι παταγώδη η αποτυχία του, στη Γαλλία τουλάχιστον γιατί οι διαρθρωτικές προσπάθειες και τα επενδυτικά ταμεία τίποτα δεν έχουν κάνει, ούτε θέσει εργασίας δημιούργησαν, ούτε την οικονομική ανάπτυξη βοήθησαν. Και μάλιστα ο Δημοτικό Σύμβουλο το διαπιστώνω αυτό καθημερινά. Απλώς κατασπαταλούμε κονδύλια σε, σε περιφερειακό επίπεδο και τίποτα, κανένα πρόβλημα δεν επιλύουμε. Υπάρχουν μεγάλες ε, ανισότητες ε, σε, στις γαλλικές περιφέρειες μεταξύ της υπαίθρου και των αστικών κέντρων και κάθε χρόνο αυξάνονται αυτές οι διαφορές. Και μάλιστα ε, η κατάσταση είναι χειρότερη για τις ε, απομονωμένες αγροτικές περιοχές ε, για να μην μιλήσουμε για την ελάχιστη πρόσβαση που έχουν σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έτσι ζουν ένα αργό θάνατο αυτές οι αγροτικές περιοχές, ενώ στο παρελθόν ήταν κινητήρη μοχλή της οικονομίας. Πώς θα γίνει λοιπόν καλύτερη κατανομή της χρηματοδότησης. Πολύ φοβούμε ότι ένα τμήμα της θα πάει στους μετανάστες. Ε, τι γίνεται με την περίοδο 2007-2013 είστε σε θέση να κάνετε έναν απολογισμό της προηγούμενης ε, προγραμματικής περίοδου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλκάρσελ Σίσο, ο αντιπρόεδρος μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και θα έχει κέρια σημασία και στο μέλλον κατά τη χρησιμοποίηση αυτών των, διαρθρωτικών, των κονδυλίων των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Επίσης, ε, καλό θα ήταν να τονίσουμε τις συνέργειες ε, και τους μηχανισμούς για το συνδυασμό των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και να αξιοποιήσουμε αυτές τις συνέργειες και στη γεωργία. Σίγουρα απαραίτητος πυλώνας είναι η καινοτομία, ο νεοτερισμός. Έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την αγροεπιστήστικη παραγωγή, να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και επίση να ενισχύσουμε την διασυνδεσιμότητα των αγροτικών περιοχών και τη υπαίθρου. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στην υπαίθρο και αυτή την άποψη η ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην καινοτομία και ε, είναι απαραίτητη και αναπόδραστη υποχρέωσή μας. Επίσης, ζωτική σημασία έχει η ενίσχυση και τη εργασία και τη απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, είτε μέσω τη καινοτομία, είτε μέσω ενισχύσεων για την ε, ε, δημιουργία επιχειρήσεων. Επίσης, σημαντική είναι και μια εκστρατεία προώθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δοθούν πληροφορίε για τι χρηματοδότικέ δυνατότητε που δίνουν τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρέπει να γίνει καλύτερη προβολή όλων αυτών των ευκαιριών και δυνατοτήτων. Και επίση ε, και οι εθνικέ αρχέ θα πρέπει να προωθούν και να εξηγούν το τεράστιο δυναμικό ε, που έχουν για την Ήπεθρο και τι αγροτικέ περιοχέ ε, τα ταμεία αυτά διαρθρωτικά και επενδυτικά. Ευχαριστώ. Κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίασή της και την εισηγήτρια για τη δική της παρουσίαση. Είναι κρίσιμο σημασία ε, να έχουμε στο μυαλό μας οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ε, στην, σε αγροτικές περιοχές. Ε, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην οποία συμμετέχω, πάρα πολύ Ανησυχούμε και προσπαθούμε να βρούμε τα εργαλεία που θα βοηθήσουν να βρεθούν θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν οι, περιοχές, οι αγροτικές περιοχές. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι στις συζητήσεις τώρα πρέπει να μπει και το θέμα της εμπλοκής των κρατικών αρχών. Δεν είναι φυσιολογικό εμείς ε, στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο να έχουμε μια σειρά αιρεσιμοτήτων και τα κράτη τελικά να βάζουν άλλους 20 με 30 όρους για να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα σας δώσω κάποια ε, παραδείγματα από τη δική μου χώρα. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν ε, εισάγει προ... περιορισμούς για το ποιος ε, μπορεί να έχει πρόσβαση στα κονδύλια, η Ρουμανία έχει πει ότι αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι κοινότητε που, που έχουν πάνω από 2.000 κατοίκους, άρα εξαιρούν κάποιους. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποδεχτούμε τέτοια μέτρα από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα των κρατών μέλων να εισάγουν πρόσθετους όρους. Ωραία, δεν βλέπω να ζητάει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα παρακαλούσα τη συντάκτρια γνωμοδότησης να αναφέρει στη γνωμοδότησή της και το πρόβλημα του ύψου ε, των κονδυλίων, των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων ε, ε, και το πώς θα διανεμηθούν αυτή στην στιγμή προκειμένου να διασφαλιστεί η εδαφική συνοχή. Γιατί δίνεται μερικέ φορές η εντύπωση ότι η η Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη δίνει περισσότερη έμφαση στις πόλεις και όχι τόσο στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε την ανάγκη να στηρίξουμε ε, και την ανάπτυξη της Ήπεθρο και να μην αμελούμε τις αγροτικές περιοχές. Γιατί στην Ήπεθρο έχουμε τις περισσότερες περιβαλλοντικές συνέπειες και εκεί χρειάζεται εξυγχρονισμός και καινοτομία στη γεωργία. Ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru comentariile tuturor uh, colegilor, precum... Στο πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και για τη συνολική παρουσίαση από την Επιτροπή. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να συνεισφέρουμε σημαντικά με την εμπειρογνωμοσύνη μας σε αυτή την έκθεση μέσα από το φίλτρο των ε, τοπικών και ε, εθνικών εμπειριών που έχουμε καταφέρει να συσσωρεύσουμε. Θα περιλάβω όσο περισσότερες συστάσεις μπορώ ε, στη γνωμοδότηση, αλλά δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλονται λόγω του μεγέθους της γνωμοδότησης, κάποιες θα πρέπει να μπουν ως τροπολογίες. Να σας πω λίγο ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Η παρουσίαση στην Επιτροπή είναι στις 30 Αυγούστου. Κατανοώ λοιπόν ότι ε, τέλη Νοεμβρίου θα είναι η <clears throat> ημερομηνία για τις τροπολογίες. Επίσης θα υπάρξει δημόσια κρόαση στην Επιτροπή Ρέτζη στις 15 Ιουνίου. Για το θέμα αυτό τι θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη γνωμοδότησή μας. Σας ευχαριστώ και περιμένω τη συνεισφορά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι η εξέταση της, ε, του σχέδιου γνωμοδότησης έγινε 30 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου 2016 γίνεται λίγη προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και η έγκριση θα γίνει 12-13 Οκτωβρίου μετά τις θερινές διακοπές. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα συμμετοχή στην ε, ε, Επιτροπή Γεωργίας του κ. Μάνια που είναι παρατηρητής από το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας. Ήταν μαζί μας ε, στην Επιτροπή Γεωργίας από το 1998. Οπότε είδε πολλούς ευρωβουλευτές που πέρασαν από αυτή την Επιτροπή. Έχει μακροχρόνια πείρα σε αυτή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγει στη σύνταξη, την αξίζει άλλωστε. Βέβαια οι υποχαιρετισμοί έχουν πάντα μια νότα θλίψης, αλλά θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά ε, τον συνάδελφο, να τον αποχαιρετήσουμε με χαμόγελο, να τον ευχαριστήσουμε για την ε, συμβολή του, τη συνεισφορά του, τη συνεργασία μας, να του ευχηθούμε καλή τύχη ε, σε ό,τι θα θα κάνει από εδώ και πέρα. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα εγκαταλείψει ε, τη Γεωργία, γιατί όσοι έχουν κάποια επαφή με τη Γεωργία και τους Γεωργούς ε, μένουν πιστοί ε, και προσιλωμένοι σε αυτούς μέχρι τέλους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Σιεκέρσκι, γιατί όχι από το 98, από το 95 είμαι εδώ και πρώτη φορά από τότε έχω την ευκαιρία να λάβω το λόγο στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θυμάμαι την πρώτη συνεδριαστή παρθενική μου συμμετοχή στην Επιτροπή Γεωργίας τότε ήταν πολύ διαφορετικό ο κόσμο και τη κοινή γεωρική πολιτική, που τότε η κοινή γεωρική πολιτική δεν ενέπιπτε στη διαδικασία συναπόφαση, γιατί τότε είχαμε ε, ε, επίπεδο, ε, ποσοστό αγρανάπαυση 5,5% επί επιτρόπου Φίσλερ. Τώρα έχουμε τελείω διαφορετικό τοπίο στη Γεωργία, τελείω διαφορετικό κόσμο στη Γεωργία, τελείω διαφορετική κοινή γεωργική πολιτική και πραγματικά είχα την τύχη να είμαι μάρτυρα ε, σε όλη αυτή τη μεγάλη περιπέτεια και αναζήτηση τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά και για την ε, βοηθεία και την στήριξη που είχα από το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας. Σας ευχαριστούμε και πάλι και όλες αυτές τις γνώσεις σας, τις εμπειρίες σας, τις παρατηρήσεις σας, καλό θα ήταν να τις αποτυπώσετε και σε ένα κείμενο για να τις αξιοποιήσουμε και εμείς και η διαδοχή μας. Νομίζω ότι είναι πολύτιμη αυτή η πείρα που συγκεντρώσατε όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια εξιστόρηση όλων αυτών των ε, εμπειριών και πολύ χρήσιμο και συναρπαστικό ανάγνωσμα για όσους ασχολούνται με τη γεωργία. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 7, τη βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Πρόκειται για ένα κανονισμό για τον οποίο η συγητής μας είναι ο κύριος Μάρτιν Χόισλινγκ, πολύ σημαντικός κανονισμός και δύσκολος, αλλά απαραίτητο. Γίνονται διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τριμέρους διαλόγου, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο αρμόδιος, ο εισηγητής μας, ο κύριος Μάρτιν Χόισλινγκ. Ε, Φαντάζομαι και ήδη βλέπω πολλοί ότι θέλουν το λόγο, αλλά ένα λεπτό θα έχει ο καθένα μετά για τι ερωτήσει του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Να πω ότι δεν θα γίνει κάποια συζήτηση βάσης ε, γιατί δεν έχει ε, ψηφιστεί ακόμα Εγώ προσπαθώ να περάσω τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου, αυτά που έχουμε αποφασίσει με μεγάλη πλειοψηφία. Ο Επίτροπος είπε και για τα βιολογικά ζητήματα ε, και στην ε, ομιλία του, είπε ότι ε, σε πολλά σημεία υπάρχουν οι ανάγκη για προτάσεις συμβιβαστικές οι οποίες ε, αποδεικνύονται δύσκολες γιατί τα τρία όργανα δεν μπορούν να έρθουν σε μια κοινή ε, θέση εύκολα, τουλάχιστον από την πλευρά της Κομισιόν. Περιμένουμε απλώς στα σημεία που ήδη υπάρχουν συμβιβασμοί να... Δεν υπάρχει μετάφραση. Υπάρχει πρόβλημα με τη δεμήνη από ποια γλώσσα. Α, αγγλικά. Δεν είχαμε αγγλική διερμηνία. Κύριε Χόσλινγκ, ίσως πρέπει να ξαναρχίσετε. Την αρχή. Να πω απλώς ότι ε, ότι για να μπορέσουν τα τρία θεσμικά όργανα να ε, συμφωνήσουν θα πρέπει να πάρουμε τις μεγάλ, τη μεγάλο αριθμό συμβασμών από την Κομισιόν. Είμαι αισιόδοξο ότι στις επόμενες διαπραγματεύσεις ε, θα πάμε ένα βήμα μπροστά. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που το λέω ξεκάθαρα, είναι ότι το Συμβούλιο δεν έχει αλλάξει ε, η εντολή του για τις διαπραγματεύσεις και αυτό είναι δύσκολο να οδηγήσει σε ενιαία θέση σε πολλά ζητήματα. Ε, όπως για το βασικό ε, κανονισμό, για την ακτινοτροφία που ε, χρειάζεται ένας τέτοιος ε, κανονισμός. Αν δεν έχει συζητήσει το θέμα αυτό το Συμβούλιο, δεν έχει εντολή και είναι δύσκολο. Επίσης, η ευελιξία από την πλευρά του Συμβουλίου, ε, αν πάει λίγο μπροστά, καλό θα ήταν, όμως πιέζει ο χρόνος και δεν γίνεται κάτι. Επίσης... ένα βασικό αίτημα ε, ε, το Κοινοβουλίο ήταν να παραμένουν οι έλεγχοι για τα βιολογικά προϊόντα. Έχουμε εδώ μια εντολή για διαπραγματεύσεις ε, που πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μια κοινή εντολή από τις Επιτροπές ΕΜΒΙ και ΑΓΡΙ που θα μπορούσε να μας πάει παραπέρα για να παραμείνουν τα βασικά στοιχεία ε, των ελέγχων ε, στον κανονισμό για τα βιολογικά προϊόντα. Είμαι αισιόδοξο ότι και σε αυτό το σημείο θα μπορέσουμε να έχουμε ε, συνεννόηση. Ένα άλλο θέμα είναι η κατεξουσιοδότηση και οι εφαρμοστικές πράξεις, ένα θέμα που υπάρχουν διαφωνίες εδώ ε, μιλάμε για τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους. Έχουμε πάει κάπως μπροστά για τα πιστοποιητικά. Ε, να πω ότι ε, και για τις εισαγωγές έχει υπάρξει συζήτηση. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους κανόνες για τις ομάδες επιχειρήσεων οι οποίες θίγονται σε, ε, στο διηνικές. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρος κανένας για την σήμανση και βέβαια ένα άλλο ανοιχτό θέμα είναι ε, πώς ακριβώς η Κομισόν θα συνεννοηθεί με τα κράτη-μέλη για να οριστεί αυτό το ε, θέμα πιο συγκεκριμένα. Υπάρχουν ε, κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μετατροπή τα οποία έχουν να κάνουν με διαφωνίες μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Επίσης, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το άρθρο 20. Εκεί είναι η αρχή πρόληψης, ε, ε, είναι ειδικά η επιβάρυνση με λιπάσματα ε, του εδάφους από την πλευρά του Κοινοβουλίου Συμβουλίου και Κομισιόν ε, υπάρχουν διαφωνίες. Ε, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο είναι σχετικά κοντά γιατί δεν θέλουμε εμείς από το Κοινοβούλιο κάποια νέα όρια, θέλουμε να αποφύγουμε απλώς αυτές οι εγκαθαρσίες να μπουν στην οικολογική παραγωγή, να μην είναι επιβαρημένοι, να μην επηρεαστεί. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει στις διαπραγματεύσεις ότι αυτό είναι ε, καθήκον και των παραγωγών και των επιθεωρητών. Να είμαι όμως αισιόδοξη ότι θα συμφωνήσουμε και σε αυτό το θέμα. Επίσης, την Πέμπτη θα ε, κάνουμε μια τρομερή διάλογο, όπως και τις επόμενες εβδομάδες. Ε, πιστεύω ότι θα πάμε μπροστά. Θα το δείξει βέβαια ο χρόνος. Βέβαια στην τρέχουσα προεδρία δεν μπορέσαμε να βρούμε ε, μια νέα θέαση. Ελπίζουμε να μην υπάρξει τίμημα για αυτό που από κοινού θα αποφασίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Εραντ Καρσία πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Ένα συγκεκριμένο θέμα ήθελα να θίξω. Τις περιοχές, τις εξόχους απόκεντρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τρίτες χώρες και τις εισαγωγές από αυτές. Αυτό που θα ήθελα είναι να προσπιστούμε τη θέση που οι ε, προσπιζόμασταν στην Επιτροπή Γεωργίας. Όταν αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός, να μπορέσουν να έχουν τις ίδιες εξαιρέσεις που προβλέπονταν και για τις τρίτες χώρες. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοια μεταχείριση κατά και ει βάρο αυτών των εξόχως από περιοχών, ενώ έχουν την ίδια γεωγραφική απόσταση με τρίτες χώρε. Οι περιοχέ αυτέ. διέπονται από άλλους κανόνες και διατάξεις σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι τρίτες χώρες θα πρέπει να επωφεληθούν από μικρότερες απαιτήσει για την πρώτη πενταετία, αρκεί να προβλεφθεί το ίδιο και για τις από απόκεντρες περιοχές. Δηλαδή θα έχουμε σοβαρή διακριτική μεταχείριση. Αυτό και πιστεύω ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να λάβει υπόψη το άρθρο 28 του κανονισμού και να προσπίσει την εντολή της Επιτροπής Γεωργίας στον τριμερή διάλογο. Η κυρία Γκέρινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, δεν έβαλα την πινακίδα μου πρώτα. Με συγχωρείτε. Άκουσα την παρουσίαση του κ. Χόισλινγκ και αυτό που είχα να πω το λέω ως εισηγήτρια, ισκαιώδης μάλλον εισηγήτρια, για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Πρέπει να δηλώσω ότι είμαι ιδιαίτερα απεσιόδοξη. Για να μην πω ότι έχω απελπιστεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Αυτό ο τριμερή διάλογο έχει κρατήσει ένα εξάμεινο πλέον. 15 ώρε συνεδρία την εβδομάδα έχουμε. Και τεχνικέ και σκιωδών. Και δεν έχουμε πετύχει και πολλά, πρέπει να πω. Πολύ λίγα έχουμε να επιδείξουμε σε αποτέλεσμα για, τέση, για τόση προσπάθεια και τόσο κόπο. Δεν έχουμε συμφωνήσει για τους ελέγχους, για τα ζεζανιοκτώνα, για τίποτε από τους κανόνες συγκεκριμένων παραγωγών. Και αυτό οφείλεται εν μέρη στο υπερπολύπλοκο και πολύ συχνά θα έλεγα ασυνεπές ε, στην υπερπερίπλοκη και ασυνεπή εντολή που είχαμε για τις διαπραγματεύσεις. Είναι από του χειρότερου τριμερεί διαλόγου του οποίου συμμετείχα ποτέ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν με εκπλήσει λοιπόν που έχουμε και τώρα δυσκολίε. Παρ' όλα αυτά κάτι πρέπει να κάνουμε και να προχωρήσουμε. Θα ε, αδράξω λοιπόν αυτή την ευκαιρία για να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων ε, στην περίπτωση των ζωνιακτών λόγου χάρη. Κάτι πως τώρα έχει παραγνωριστεί. Ο εισηγητής έχει πλήρη προθυμία να προστατεύσει το εμπόριο και την ε, ε, παραγωγή της βιολογικής γεωργίας, του οποίου τυχαν είναι και μέλος και ενδιαφερόμενος, εις βάρος των καταναλωτών. Αυτό νομίζω ότι έκανε όταν ε, οργάνωσε την ψηφοφορία. Με τη θέση που προωθεί, οι γεωργοί θα μπορούν να θέτουν στην αγορά για εμπορία προϊόντα που θα παρουσιάζονται ως βιολογικά, ακόμη και αν έχουν μολυνθεί από ζυζανιοκτώνα, όπω και τα κλασικά προϊόντα, τα παραδοσιακά. Αυτό δεν τον πειράζει, δεν πειράζει για του γεωργού, αλλά αναρωτιέμαι τι γίνεται για του Με του καταναλωτέ. Εγώ αγοράζω βιολογικά προϊόντα και δεν θα ήθελα να έχουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων ή ζυζανιοκτώνων όταν τα κατάλληλα λοιπόν, αυτήν την άγουσα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Η ζυζανιοκτωνα οταν τα αγοραζω δεν καταλαβαινω αυτή απλώς υπονομεύει και ε, κάνει αξιόπιστο τον όλο τομέα. Και παρόλα αυτά, μαζί με άλλα ζητήματα, ε, κάνει τι διαπραγματεύσει να χρονοτριβούν. Ρωτώ λοιπόν ξανά, γιατί παίρνει τόσο πολύ καιρό να λυθεί το ζήτημα αυτό. Έχω πάρα πάρα πάρα πολλά νομοθετήματα πίσω μου στην εμπειρία μου και δεν θα εδώ για να σπαταλάω το χρόνο μου. Έχω πολλέ υποχρεώσει ω κοιόδη ε, εκ μέρου τη ομάδα μου και πραγματικά εδώ έχουμε χαλάσει πάρα πολύ χρόνο. Ε, θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν τον συγητή λιγάκι να ανασκουμποθεί, να επιταχύνει και εντάξει δεν είναι πολύ διαλλακτική το Συμβούλιο, αλλά ούτε εκείνο είναι διαλλακτικό. Οι διαπραγματεύσει ε, ε, προποθέτουν κινήσει και από τι δύο πλευρέ. Καμία συμβαστική διάθεση δεν βλέπουμε από πλευρά του. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνει και να προχωρήσει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε διαρκώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βιαστούμε στην ψηφοφορία για να προλάβουμε στην Προεδρία του Λουξεμβούργου. Έτσι είχαμε πει και τελικά έχουμε φτάσει στο τέλο τη Ολλανδική Προεδρία. Τελειώνει και αυτή. Τι να πω. Πραγματικά δεν θέλω να είμαι δυσάρεστη. Ελπίζω να μην είμαι αγενή, αλλά έχω φτάσει στο σημείο που βρίσκω ότι είναι ένα φρικτό αστείο όλο αυτό. Και δεν καταφέρνουμε και τίποτα. Πολύ δυνατά τα λόγια σα. Κύριε Κέστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος ε, Χόισλινγκ ε, ανέφερε ένα πολύ πιεσμένο χρονοδιάγραμμα. Ε, όταν μιλάμε για τη φυτοπροστασία και τα φυτοπροστατευτικά μέσα, η συζήτηση είναι πάρα πολύ και έντονη και αυτό έχει να κάνει και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχουμε κλειστά συστήματα ε, για την παραγωγή αυτών των προϊόντων, έχουν με εξωτερικές επιρροές. Ειδικά η συζήτηση για τα κοινά όρια. Υπάρχει δυνατότητα τελικά να καταλήξει με καλό τρόπο όπως και στο παρελθόν ε, υπάρχει η δυνατότητα το κάθε κράτος μέλος ε, να δώσει τα δικά του όρια. Αυτό θα το διατηρήσουμε. Ε, πάρα πολλά κράτη-μέλη θεωρούν αυτό δεν έχει νόημα. Και κάνουν έκκληση στον εισηγητή να επηράσει μαζικά και να εκπροσωπήσει τη θέση μας. Το θέμα που σχετίζεται με όλα αυτά είναι το θέμα της ευθύνης ε, συγκεκριμένα. Ε, ποιος θα ευθύνεται για την ε, επιμόλυνση των προϊόντων είναι κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί ξεκάθαρα. Δεν πρέπει να έχουμε ανασφάλεια δικαίου για τους παραγωγού βιολογικών ε, προϊόντων και πρέπει αυτή την υποχρέωση να την αναλάβει ο εισηγητή. Επίσης, έχω ένα ερώτημα για το θέμα των σπόρων. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, οι σπόροι δεν έχει να κάνει με τους μεγάλους ομίλους στο θέμα των βιολογικών προϊόντων. Ε, ε, κατά πόσο υπάρχει πρόοδος ε, ως προς το προβάδισμα ποιότητας που έχουμε στην παραγωγή σπόρων βιολογικών. Θέλουμε να πούμε, θέλω να πω ότι έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν σπόρους οι οποίες περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία να ε, οριστεί το θέμα για να αγοράζει ο, κόσμος από αυτούς και όχι από πολυεθνικές. Θα πρέπει ο εισηγητής να αναλάβει την ευθύνη να κάνει κάτι και για αυτόν τον τομέα. Δύο λεπτά. Λίντς. Πολύ σύντομα θέλω ε, να πω κάτι σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκέρλινγκ ε, στο τριμερή διάλογο. Ε, επειδή συμμετέχω και εγώ, έχω μια άλλη αντίληψη. Από τη μία είναι σωστό ότι όντως πάμε ε, σημειωτών, όμως θεωρώ ότι η στάση του συναδέλφου Χόισλινγκ ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία ε, θυμίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε αυτό τον τριμερή διάλογο. Εμείς ως Κοινοβούλιο και Συμβούλιο έχουμε για παράδειγμα ε, μια κοινή θέση. Δεν είναι ευθύνη της Κομισιόν σε διάφορες μορφές να φέρνει εκδοχές των ορίων μέσα από διάφορα άρθρα γιατί αυτό κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά και ε, πρέπει εξ αρχής να συζητήσουμε εάν θέλουμε μέχρι τον Νοέμβριο και ως Κοινοβούλιο και ως Συμβούλιο να έχουμε αποφασίσει πολιτικά αυτό το θέμα. Μπορεί να μην ε, γίνεται με άλλο τρόπο, αλλά πολιτικό, ε, πολιτικός δεν είναι σωστή η στάση της Κομισιόν σε αυτό το θέμα ειδικά. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χόισλιν και εγώ. Άκουσα ότι υπερασπίζεστε στεναρά τη θέση του Κοινοβουλίου και εμείς ως Σκανδιναβοί και μάλιστα Φινλανδοί έχουμε Έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσει. Θέλουμε την πιο αγνή βιολογική παραγωγή, όπως την έχουμε εμείς στο βορρά. Ε, βλέπω τι συμβαστικέ προτάσει προτείνονται και δυστυχώ το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν είχαν αρκετά καλή βούληση ω τώρα. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την καλή βούληση να τη βρούμε για να μπορέσουμε αυτά τα ζητήματα να τα επιλύσουμε. Θα πρέπει να σα ευχηθώ κάθε καλή τύχη σε αυτόν τον αγώνα ώστε ο Βορρά της Ευρώπης να διατηρήσει και την καθαρή βιολογική του παραγωγή. Ευχαριστούμε κύριο Λουαζό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε η Γαλλία είναι η τρίτη παραγωγός βιολογικών προϊόντων μετά την Ισπανία και την Ιταλία. Μάλλον ε, μετά την Ισπανία και την Ιταλία και πριν τη Γερμανία. 10% αύξηση από το 2014 και 60.000 ε, θέσεις εργασίας άμεσες και πλήρους ε, χρόνο απασχόλησης. Θέλουμε λοιπόν η βιολογική παραγωγή να είναι μέρος του γεωργικού τομέα και η Γαλλία να αποφεληθεί από έναν τρόπο διατροφής που ολοένα και βελτιώνεται. Οι καταναλωτές όμως όπως ξέρετε έχουν λίγο ε, απελπιστεί με αυτά τα επαναλημμένα σκάνδαλα, τα, τα διαρκή σκάνδαλα για την τροφική της τροφικής αλυσίδας. Θα πρέπει τα σήματα των βιολογικών προϊόντων να αποδίδονται αυστηρά. Όχι απλώς να πουλούνται κάποια πράγματα ακριβότερα ή οποροκυπευτικά που πουλούνται ασχέτως ε, εποχιακής διάθεσης από χώρες που έχουν προδιαγραφές πολύ χαλαρότερες από την Ευρώπη και που μπορεί επίσης να προκαλούν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω της μεταφοράς του από αλλού. Ένα φρούτο βιολογικό ε, ε, που έρχεται ε, από χώρα από την οποία μεταφέρεται με αεροπλάνο παράγει 10 20% περισσότερο αέρα του θερμοκηπίου από ένα προϊόν που καταναλώνεται στην σωστή εποχή. Πρέπει λοιπόν να πράγουμε τα προϊόντα των τοπικών καλλιεργειών με τους σωστούς κανόνες βιολογικής καλλιέργειας. Δεν είναι θέμα μόδας ούτε δόγματος η βιολογική παραγωγή. Έχει να κάνει με την ε, διαφορετική πρακτική σε σχέση με τη βιομηχανοποιημένη γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν την οικολογική παραγωγή να την προσπιστούμε και το ίδιο για το τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε τις διατρεφικές ε, συνήθειες που θα ενισχύσουν και τις ανάγκες των γεωργών μας και τις δικές μας προσδοκίες περί ποιότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Άγγενιου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ενημερωθώ είτε από την Επιτροπή είτε από τον κύριο Χόισλιν και δύο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την βιολογική γεωργία. Γιατί έχω υποστεί πολλές πιέσεις και λόμπι. Ε, ο συνάδελφος από τη Σκανδιναβία δεν αναφέρεται. ότι πρόκειται για καλλιεργητούς σαλάτας που πλησιάζουν κοντά στον ε, αρκτικό κύκλο που δεν, δεν ε, ε, καλλιεργούν στο έδαφος γιατί είναι παγωμένο, αλλά τα βάζουν σε βαρέλια, τα βάζουν χώμα σε βαρέλια και σε θερμοκήπια. Και έμαθα ότι σταμάτησε πια αυτό ο τρόπο παραγωγή. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ενημερώσει ο συνάδελφος Τάκουλα αν υπήρχε κάποια εξέλιξη. Επίση, για του βιολογικού σπόρους Αν ο σπόρο δεν παρήχθη με τρόπο βιολογικό, τότε δεν μπορεί κανεί να το σπείρει. Είναι όμω τόσο μικρή αγορά των σπόρων που η βιολογική ε, γεωργοί θα μπορούσαν να βρεθούν είτε σε θέση που να πρέπει να χρησιμοποιούν ε, ε, σπόρους που δεν ήταν βιολογικοί ή αν χρησιμοποιούσαν σπόρους που δεν είναι βιολογικοί να μην μπορούσαν να πουλήσουν τα προϊόντα ως βιολογικά ακόμη και αν τα καλλιεργούσαν με βιολογικό τρόπο. Υπήρξε κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων γιατί η βιολογική παραγωγή μπορούν να χρησιμοποιήσουν ροτενών που είναι ένα δυσάρεστο με δυσάρεστη δραστική ουσία, αλλά είναι βιολογική. Ε, τα κατάλοιπα αφορούν και τη ροτανόνη που είναι βιολογικό, βιολογική ουσία ή μόνο αφορούν τα συνθετικά φυτοφάρμακα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αρχικά δεν ήθελα να ζητήσω το λόγο, αλλά άρχισε να με προβληματίζει και να με ανησυχεί αυτή η συζήτηση δυνατότητα δηλαδή να επιτρέψουμε ε, ή μάλλον να έχουμε κατάσταση όπου βιολογικά προϊόντα έχουν ε, μολυνθεί τυχαία, επιμολυνθεί τυχαία από φυτοφάρμακα. Γι' αυτό δεν ευθύνεται ο Γεωργός. Δεν ήταν δική του επιλογή αυτή η μαλλον να εχουμε κατασταση οπου βιολογικα προιοντα εχουν μολυνθει τυχαια επιμολυνθει τυχαια απο φυτοφαρμακα γι αυτο δεν ευθυνεται ο γιωργος δεν ηταν δικη του επιλογη αυτη η επιμολυση Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε την θέση εμπορία αυτών των προϊόντων βιολογικών γιατί αυτό θα ήταν παραπλανητικό από τη στιγμή που φέρουν και κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι και πιο ακριβά από τα συμβατικά. Θα ήταν άδικο λοιπόν για τον καταναλωτή και παραπλανητικό. Θα πρέπει να προσέξουμε και να φροντίσουμε ε, ίσως η Γεωργή να συνάπτουν ασφαλιστικά συμβόλαια ώστε να προστατεύονται και από τις επιμολύσεις όπως προστατεύονται από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Εγώ δεν συμφωνώ να έχουμε διαφορετικά επίπεδα για παρόμοια προϊόντα, ε, διαφορετικά επίπεδα δηλαδή για παρόμοια προϊόντα σε διάφορες χώρες. Θα πρέπει τα ίδια κατόφλια ε, να ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιολογικά προϊόντα. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά έχετε το πολύ, κύριε Χόισλινγκ. Äh, Ευχαριστώ να μιλήσω για κάποια θέματα που, για τα οποία έδωσα, έγιναν ερωτήσεις. Για, τις, ε, για τους χώρους κοινοτροφίας στις βόρειες ε, ε, χώρες. Να πω ότι κάθε παραγωγή πρέπει να είναι βιολογική. Δεν υπάρχει μια εξαίρεση για τις βόρειες χώρες σε αυτόν τον κανονισμό και σύμφωνα με την εντολή μας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είχα προσφέρει ένα συμβιβασμό με τον οποίο οι συνάλφοι από τη Φιλανδία και τη Σουηδία μπορούσαν να ζήσουν ε, ε, οι χώρες αυτές ε, να ξεκινήσουν άμεσα την παραγωγή με αυτό το συμβιβασμό. Όμως, ε, για, από, οι αρχές της βιολογικής παραγωγής ε, είναι πολύ μακριά από αυτό. Σε άλλες χώρες δεν αντιστοιχούν με τις βασικές αρχές της βιολογικής παραγωγής, οπότε ε, δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα συμβιβασμό. Ε, θα πάμε ένα βαθμό πάνω από ό,τι φαίνεται από τη συζήτηση. Για το θέμα των σπόρων είναι ένα θέμα που είχαμε ξεκάθαρη εντολή, τι χρειάζεται ο οικολογικός τομέας, χρειαζόμαστε οικολογικούς ε, σπόρους, όμως όταν μιλάμε για το στάτους αυτό θα πρέπει κανείς να προσπαθήσει η σκληρά να μην το χάσει. Πρέπει να είμαστε πολλές φορές βέβαια πιο ευέλικτοι γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η αγορά και να, ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς να αναπτύσσονται και οι ορισμοί. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα ορίσουμε τον, τους οικολογικούς σπόρους. Έχουμε μία ε, στον δικό μας, έναν ορισμό στον δικό μας κανονισμό ε, μετά η Κομισιόν βέβαια λέει ότι πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό βάσει της εντολής του Συμβουλίου για να προχωρήσει το θέμα. Όμως δεν είναι και τόσο απλό, διότι λέμε ότι απαιτούμε σε 10 χρόνια όλοι οι καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων να έχουν βιολογικούς πόρους. όμως η κατάσταση σε κάθε χώρα είναι διαφορετική, η αγορά θα εξελιχθεί διαφορετικά, πρέπει να αντικατοπτρίσουμε αυτή την εξέλιξη. Ένα άλλο αμφισβητούμενο θέμα είναι οι οριακές ε, τιμές. Ε, έχουμε ένα ξεκάθαρο, στο ε, Κοινοβούλιο ξεκάθαρη εντολή, διότι υπάρχουν διάφορες αξιολογήσεις και υπάρχει και μία επιβάρυνση και δεν μπορούμε να περιμένουμε από, τους, τα βιολογικά προϊόντα να ζούμε σε έναν παράλληλο κόσμο και να λέμε ότι δεν πρέπει να ε, περιλαμβάνουν καθόλου λιπάσματα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ε, πρέπει ο κανονισμός να είναι ξεκάθαρος. Είναι κάτι αναπόφευκτο αυτή η επιβάρυνση ή όχι. Και αν υπάρξει ξεκάθαρος κανονισμός ε, θα μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έχει κατατεθεί πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση για να ενισχύσουμε το τομέα αυτό. Ε, οι γεωργοί θέλουν να μεταθέσουν την ευθύνη και αυτό το σημείο πραγματικά είναι αποφασιστικό και πολύ ευαίσθητο φυσικά. Κυρία Γκέρλινγκ, θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο να λέτε ότι ο τρόπος που γίνονται οι διαπραγματεύσεις ευθύνεται για, την, ε, για το γεγονός ότι δεν πάνε μπροστά. Όπως σας είπε και ο σκιώδης εισηγητής, όλα τα έχουμε εκ των προτέρων συμφωνήσει με τους Σκιώδης εισηγητές και όταν πρόκειται για συμβιβασμούς τους έχουμε συμφωνήσει και για τα τεχνικά μέσα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ε, δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι αν θέλουμε αν το κάνουμε λίγο διαφορετικά, να δούμε τι θα κάνατε τότε κυρία Γκέρλινγκ, αν έπρεπε όλοι να συμμετέχουν θα ήταν πάρα πολύ δουλειά. Ναι, είναι πολλή δουλειά, αλλά δεν μπορούμε και γρήγορα να αποδώσουμε, αν θέλουμε να αποδώσουμε σωστά. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω πιο γρήγορα γιατί πρέπει να τηρήσω αυτά που έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι η δική σας ομάδα δεν ε, συμφωνεί με πολλά από αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Όμως πρέπει να τα αποδεχτείτε και να αφήσετε τα πράγματα να εξελιχθούν. Δυστυχώς, αν είναι κακή η εντολή διαπραγματεύσεων, ε, δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν είναι δημοκρατικό όταν το έχει αποφασίσει η μεγαλύτερη πλειοψηφία. Πρέπει να το αποδεχτείτε και να πείτε ότι αυτό είναι η ιδιωτική γνώμη σας και όχι αυτή ε, του Κοινοβουλίου, όταν εσείς έχετε διαφορετική γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χόισλινγκ. Έχουμε διεκπαιρεώσει τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Μην ξεχνάτε αύριο την ακρόση που θα έχουμε για το γάλα. Θα ξεκινήσει στις 7 ε, και θα κρατήσει μέχρι τις 10.30. Ε, μέχρι τις 10, συγγνώμη. Όχι 9.30 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά 7 με 10. Μην ξεχνάτε την αυριανή δημόσια κρόση, που θα είναι εκτενής δημόσια κρόση, για το γάλα επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 6 Ιουνίου, αλλά ούτως ή άλλως θα τα πούμε και αύριο. Στη σημαντική αυτή ακρόαση για το γάλα που ελπίζω να είμαστε όλοι παρόντες. Σας ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση. Καλό απόγευμα.